Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ξεκινάμε σήμερα την δεύτερη συνεδρίασή μας, η οποία θα αφιερωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013, που είχε ως κεντρικό του θέμα την άμυνα Πρέπει να σας πω ότι με την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με την κυρία Αρνό και τον πτέραρχο Ρουσιέ θα καλύψουμε όλο το πρώτο τμήμα της πρωινής συνεδρίασης και θα συνεδριάσουμε από κοινού και με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά την έκθεση για την γενική σφαιρική προσέγγιση. Πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω την έκθεση αυτή με την ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ και θα αφιερώσουμε το τελευταίο τμήμα της πρωινής μας συνεδρίασης 12 με 12.30 ακριβώς στην ε, συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε πάντως πολύ γρήγορα γιατί τόσο άλλως υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία για την έκθεση αυτή. Πριν από μερικές μέρες ξεκινήσαμε λοιπόν συζητήσεις με εκπροσώπους από διάφορα όργανα στα οποία δόθηκε εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν τα συμπεράσματά του. Ε, συζητήσαμε τον κύριο Σερανό από το Συμβούλιο, τον κύριο Ποπόφσκι και έχουμε σήμερα μαζί μας δύο σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει φαντάζομαι θα πούνε το αντίθετο να είναι ικανοποιημένοι με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μόλον ότι γνωρίζουν ότι εμεί ω ευρωβουλευτέ έχουμε κάποιε επιφυλάξει και κάποιου ενδιασμού σε σχέση με την έλλειψη ενός υψηλού βαθμού φιλοδοξίας στα συμπεράσματα αυτά. Ο πτέραρχος πάντως ε, Ντερουζιέ που είναι μαζί μας τώρα και η κυρία Αρνού που θα είναι λίγο αργότερα μαζί μας, έχουν λάβει από το Συμβούλιο επισήμως έναν συγκεκριμένο σαφή οδικό χάρτη, και θεωρώ ότι και οι δύο θα πρέπει ουσιαστικά να είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα αυτό. Βέβαια εσείς επισήμως θα το πείτε αυτό. Ο πτέραρχος κύριος Ντερουζιέ, ο οποίος έρχεται συχνά στις συνεδριάσεις μας και είναι επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάνει μια παρουσίαση και έναν απολογισμό των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βέβαια κύριε Ντερουζιέ μπορείτε να αναφερθείτε και σε άλλα ζητήματα Είχαμε πριν από μερικές μέρες εδώ πέρα την ύπατη εκπρόσωπο. Μιλήσαμε επίσης για την τελευταία αυτή στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Για την αποστολή αυτή δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες ακόμα. Θα μπορούσατε ενδεχομένω εσείς λίγο να μας διαφωτίσετε. Κύριε Πτεραρχέ, μου έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντα τιμή μου να εμφανίζουμε εδώ και να απαντώ στις ερωτήσεις σας για την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Είναι πολύ χρήσιμο και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Ε, μου είπατε ότι θέλετε να σας μιλήσω για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της, ε, που έλαβε για την έρευνα, για την άμυνα, ε, το οποίο ήταν το πρώτο με παρόμοιο θέμα από το 2008. Καθώς επίσης και στη συνέχεια που θα δοθεί. Πριν όμως ε, περάσω σε αυτό, ε, θα ήθελα να σας ε, να τοποθετήσω τα λόγια μου σε ένα γενικό πλαίσιο. Όπως ξέρετε, η προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφορετικότητα και ο συνδυασμός των εργαλείων που διαθέτουμε για την επίλυση κρίσεων, περίπλογων κρίσεων. Έχουμε πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά, ανθρωπιστικά, δικαστικά, αστυνομικά και στρατιωτικά μέσα. Αυτή είναι μια συνολική προσέγγιση, πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προβλέψει ε, και να δράσει προληπτικά εναντί κρίσεων. Αυτό την καθιστά αναγνωρισμένο παίκτη στην διεθνή σκηνή. Και επίσης αυτός ο χαρακτήρας της ε, ε, την καθιστά κρίσιμη στην επίλυση διαφορών σε ζώνες που εμφανίζονται συγκρούσεις. Ε, γι' αυτό το λόγο τα 28 κράτη-μέλη δείχνουν την αλληλεγγύη τους ε, και θέτουν ε, μέσα σε κοινή διάθεση. Ε, όμως, έχουμε πολύ πρόοδο μπροστά μας να κάνουμε. Από την τελευταία φορά στην οποία σας μίλησα, πριν από ένα χρόνο, έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αρκετά σημεία. Να ξεκινήσω από τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 3.000 ε, ε, στρατιώτες υπό ευρωπαϊκή σημαία ε, που υπηρετούν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχουμε πέντε αποστολέ αυτή τη στιγμή. Πρώτον, η στρατιωτική αποστολή εκπαίδευση στο Μαλί ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2013. 23 κράτη-μέλη συμμετέχουν. Παρόλο ότι ορισμένα από αυτά δεν είχαν κανένα ιστορικό δεσμό ή πολιτικό συμφέρον συνδεόμενο με την περιοχή αυτή. Έχει ήδη πετύχει αυτή η αποστολή. 1.800 στρατιώτες του Μάλι έχουν ήδη εκπαιδευτεί και έχουν αναπτυχθεί στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ταυτόχρονα το τέταρτο τάγμα τελειώνει την εκπαίδευσή του. Τέλος, η απόφαση να παραταθεί η, απόφαση, η αποστολή μέχρι το Μάιο του 2016 λήφθη πρόσφατα ε, και από το Συμβούλιο. Θα επιτρέψει την εκπαίδευση τεσσάρων ακόμα ταγμάτων ε, και θα δώσει μια αποκεντρωμένη υποστήριξη για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Θα ε, δώσουμε βοήθεια στις αρχές του Μαλή να εξυγχρονίσουν το στράτευμα τους. Δεύτερη αποστολή, η αποστολή Αταλάντη για την καταπολέμηση πειρατείας στο κέρας της Αφρικής. Ε, από πέρσι που σας μίλησα έχει δώσει πρόσθετους καρπούς. Ε, οι επιθέσεις, οι πειρατικές επιθέσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Ε, η συνεργασία γίνεται και με, με τα άλλα σώματα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην περιοχή, Νέστορ, Στολή Νέστορ, Αποστολή, Επιχείρηση Σομαλία κλπ. Ε, όμως ε, δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε διότι οι πειρατές δεν έχουν εξαφανιστεί. Ε, γίνονται ακόμα απόπειρε ε, επιθέσεων. Τέλος, ε, ελήφθη πρόσφατα απόφαση για την παράταση της ε, επιχείρησης αυτής μέχρι το Δεκέμβριο του 2016. Τρίτη αποστολή είναι και πάλι στρατιωτική αποστολή εκπαίδευση στη Σομαλία. Και αυτή η αποστολή ε, μετακινήθηκε στο Μογκαντήσο, αυτό είναι ένα κρίσιμο στάδιο. 3.800 στρατιώτες ε, Σομαλοί εκπαιδεύτηκαν στην Ουγγάντα και πάνω από 1.000 ακόμα στρατιώτες θα ε, μεταφερθούν στην Σομαλία κατά τη διάρκεια του 2014. Μεταξύ αυτών θα εκπαιδεύσουμε εκπαιδευτές οι οποίοι αργότερα θα εκπαιδεύσουν τα δικά του στρατεύματα. Τέταρτη επιχείρηση είναι η Αλτέα. που δίνει σημαντική βοήθεια στις αρχές της Βοσνίας Αρζεγοβίνης για να ε, επιλύσουν το πρόβλημα του οπλισμού ε, ο οποίος έχει περισσέψει και αποτελεί κίνδυνο ε, για το μέλλον. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις αποφάσισε τη Δευτέρα να, να ξεκινήσει μια επιχείρηση ε, στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την U4. Ε, θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα στην περιοχή του Μπάγκη μέχρι ότου η αποστολή υποστήριξη προ την Κεντρική Αφρική υπό Αφρικανική ηγεσία να αναπτύξει τα δικά τη στρατεύματα. διορίστηκε ο επικεφαλή τη επιχείρηση, ο Φιλίπ Ποντιέ, ενώ η Ελλάδα έθεσε ε, το στρατιό της Λάρισας στη διάθεση της επιχείρησης αυτής. Όλα αυτά επιτρέπουν να αναπτυχθούν γρήγορα τα στρατεύματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Αυτή η αποστολή αυτή η επιχείρηση θα γίνει σε στενή συνεργασία προφανώ με τι ε, άλλε δεσμεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα τι ε, δεσμεύσει σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, την αναπτυξιακή βοήθεια και τέλο στο πλαίσιο τη χρημα, τη ε, της οικονομικής ενίσχυσης της αποστολής στην Αφρικανική Ένωση. Τώρα, τι έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες το τελευταίο χρόνο. Η εκτελεστική διευθύντρια της ε, υπηρεσίας, ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας θα πει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα τα πράγματα προχωράνε. Το Ευρωπαϊκό Επιτελείο Νέων Μεταφορών, για παράδειγμα, που περιλαμβάνει τον γερμανικό, ολλανδικό, βελγικό, γαλλικό και λουξεμβουριανό ε, στρατό ε, με 150 συνολικά αεροπλάνα τα οποία βασίζονται στο Eindhoven και ε, συνεργάζονται καθημερινά. Ε, το δράμα των φιλιοπινών, η επιστροφή των στρατιωτών από το Αφγανιστάν, οι καθημερινές δραστηριότητες εκπαίδευσης αυτών των πέντε χωρών, η ανάπτυξη ε, μέσων στο Μάλι και στην Κεντρική Αφρική αποτελούν ορισμένα από τα επιτεύγματα ε, αυτού του επιτελείου. Λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του. Εν τω μεταξύ έχουμε, ε, έρχονται και καινούργια μέλη. Η Ισπανία θα ενταχθεί στις 3 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Επιτελείο Νέων Μεταφορών. Αυτό αποτελεί σημάδι της σημασίας του επιτελείου αυτού. Άλλα κρατημέλη έχουν επίσης εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε αυτή τη δομή. Ορισμένα μάλιστα έχουν ε, υποβάλει και επίσημες ε, αιτήσει ένταξης. Δεν θα σας πω ποιες είναι, θα το ανακοινώσουν οι ίδιες οι χώρες. Το λέω αυτό διότι κατά την άποψή μου αυτό το παράδειγμα δείχνει ε, τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Προφανώς δεν πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό στρατό, ε, ούτε μια Ευρωπαϊκή πολεμική αεροπορία. Αλλά θέλουμε να ε, αυξήσουμε την ελεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτρέψει ε, την ανάπτυξή μας σε οποιαδήποτε πλαίσιο. Τώρα, περνάω στην προετοιμασία του Συμβουλίου. Εδώ και ένα χρόνο έγιναν πολλά πράγματα για την προετοιμασία του Συμβουλίου. Πολλοί έλεγαν ότι δεν θα καταλήξει πουθενά. Πιστεύω όμω ότι συνέβη το ακριβώ αντίθετο. Εδώ και ένα χρόνο, εδώ στι Βρυξέλλε, εγώ ήμουν μάρτυρα του πώ ε, τα 28 κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξαν δυναμισμό και η Επιτροπή σας μάλιστα ήταν ιδιαίτερα πρωταγωνιστική. Στο πλαίσιο της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής οι αρχηγοί ΓΕΣ συζήτησαν συχνά, έκαναν προτάσεις οι οποίες ε, κατευθύνθηκαν στους ε, υπουργούς και κατόπιν στους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων εν ώψη του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Τέλος, το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου επέτρεψε στους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων να συζητήσουν ε, με καρποφόρο τρόπο ε, κάτι που δεν είχε συμβεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή λοιπόν. Έχουμε ένα οδικό χάρτη, στον οποίο αναφερθήκατε εσείς πρόεδρε, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Πρώτον, Ιούνιο του 2015, για την αξιολόγηση της ε, πρόοδου και για να δώσουν καινούργιες ε, ε, κατευθύντες γραμμές οι αρχή κρατών κυβερνήσεων. Και μετά το, 2000, τον, το καλοκαίρι του 2014, μια ενδιάμεση έκθεση με την ε, δημιουργία πρόταση μιας ε, θαλάσσης στρατηγικής με συστάσεις για τη βελτίωση του equipment support, ε, τη βελτίωση της, των δυνατοτήτων αντί, ταχείας αντίδρασης Ευρωπαϊκής έκθεση για τη χρηματοδότηση των αποστολών και των επιχειρήσεων της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και τέλος της, τη μελέτη των ενωτών που έχουμε για τον έργο των σύνορων στην περιοχή της Σαχάρας και του Σαχέλ. Ε, και ε, η Στρατιωτική Επιτροπή θα έχει πολλή δουλειά να κάνει. Ε, θα σας μιλήσω για πέντε προτεραιότητες που έχουμε. Καταρχήν είναι ανάγκη να αναπτύξουμε μακροπρόθεσμα και συστηματικά τη συνεργασία στον τομέα της, του προγραμματισμού της ε, άμυνας. Μιλώ για συνεργασία, όχι κοινό σχεδιασμό. Δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε την διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για να ε, επιτρέψουμε τη σύγκληση των αναγκών σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και το συντονισμό των χρονοδιαγραμμάτων των κρατών μελών. Αυτό ασφαλώς άμεση συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Δεύτερη προτεραιότητα, ε, ε, επεξεργασία μιας στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις ε, διαστάσεις οικονομική, ανθρωπιστική, οικολογική, στρατιωτική κλπ. Ε, πρέπει να ακολουθήσουμε και να ενισχύσουμε την ανταγή προφοριών για να βελτιώσουμε την παρακολούθηση των θαλασσών. Πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια στη θάλασσα, λαμβάνοντα υπόψη την πολιτική ε, επιθυμία βούληση των κρατών μελών, ε, το ε, επιχειρησιακό, την επιχειρησιακή του τεχνογνωσία και την εμπειρία του στην κοινή δράση. Επίση, θα πρέπει να αναζητήσουμε συνέργειε ανάμεσα στο στρατιωτικό σκέλο και το πολιτικό σκέλο τη άμυνα η επιχείρηση Αταλάντη έδειξε ότι ε, λύσεις ενός θαλάσσιου προβλήματος ε, δεν είναι ούτε μόνο θαλάσσιες ούτε μόνο στρατιωτικές. Ε, τρίτο θέμα, ενίσχυση του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πολύ από τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων στο Συμβούλιο στη Συνοκορφής του Δεκεμβρίου. Με το ΝΑΤΟ συμμεριζόμαστε τις ίδιες αρχές αντιμετωπίζουμε προκλήσεις ίδιες και οι δύο οργανώσεις πολλές φορές λειτουργούν παράλληλες ίδιες ζώνες. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τον θεσμικό διάλογο με τον ΝΑΤΟ, την συνεργασία μας από την φάση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων και επίσης να ενισχύσουμε την συνέπεια ε, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ε, ε, δυνατοτήτων. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτη και από τις δύο πλευρές έτσι ώστε ε, η αντιμετώπιση μας να είναι σφαιρική. Ε, από την συνάντηση του Δεκέμβριου μέχρι τη συνοκορυφή του Νιούπορτ ε, το Σεπτέμβριο μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτά τα θέματα. Τέταρτο, τέταρτη προτεραιότητα, η βελτίωση των δυνατοτήτων ταχείας αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εδώ πρόκειται κυρίως για την ανάπτυξη της δυνατότητας ε, ε, ανάπτυξης και ευελιξίας των μάχημων μονάδων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι να δοθεί περισσότερη προσοχή στην διαδικασία λήψη αποφάσεων αλλά και στον έγκαιρο σχεδιασμό καθώς επίσης και στο θέμα της ε, χρηματοδότησης και κυρίως χρηματοδότησης ανάπτυξης ε, των στρατευμάτων. Επίσης όμως ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε και την δυνατότητα ταχείας αντίρρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά και την μεταρρύθμιση των συστημάτων ασφαλείας. Άρα λοιπόν έχουμε, πρέπει να δράσουμε και σε επίπεδο μάχημων μονάδων και σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων του τομέα ασφάλειας. Πέμπτη ε, προτεραιότητα ε, τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Η αυτοματοποίηση με ρομπότ ε, στα θέατρα της μάχης λαμβάνει χώρα σε όλους τους τομείς, στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Αυτό το ζήτημα θέτει δεοντολογικά, ηθικά ζητήματα, καθώς επίσης και ζητήματα σχετικά με το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών. Δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε από την τεχνολογία, θα πρέπει όμως να τη λάβουμε υπόψη. Ε, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Θα πρέπει λοιπόν να ε, σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε μαζί και να δώσουμε μια πολιτική απάντηση σε αυτό που ε, εγώ θεωρώ ότι είναι σημείο συνέχειας σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες. Σε, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε μαζί και μαζί και μαζί λέω. Προφανώς το κάθε κράτος μέλος θα αναπτύξει τις δυνατότητες του αυτόνομα ή επί τη βάση δημερών συμφωνιών. Ε, εμείς όμως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε μαζί πώς ε, θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μη επανδρομένα οχήματα στη στεριά θάλασσα ή τον αέρα. Αλλά νομίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να εστιάσουμε στα εναέρια οχήματα. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι πιο σημαντικές δυνατότητες. Ε, συμπληρώνουν τους ε, τις ε, πλατφόρμες αναγνώρισης και τους δορυφόρους παρακολούθησης. Έχουν τα μη επανδρομένα οχήματα, ξέρετε, έχουν αποδείξει την σημασία τους για τον εντοπισμό, την προστασία κλπ. Χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο για να καταλήξουμε ε, στην ε, δημιουργία ε, τηλεκατευθυνόμενων ενέργειων οχημάτων έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης φιλόδοξο και πολύ απαραίτητο. Καταρχήν θα έχουμε ένα πρόγραμμα για τη νέα γενιά drones αλλά και μια συνεργασία μεταξύ αυτών των χωρών που έχουν και λειτουργούν τέτοιου είδου οχήματα. Τρίτον, συνέργειε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στον ρυθμιστικό τομέα, έτσι ώστε να ενταχθούν αυτά τα οχήματα στην, ε, στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό σύστημα, αεροπορικό σύστημα. Τέλος έχουμε την χρηματοδότηση των δραστηριότητων έρευνας και ανάπτυξης. Σε στρατηγικό επίπεδο πρέπει να δούμε το θέμα της χρήσης, να δούμε το θέμα μάλλον από την πλευρά της χρήσης, έτσι ώστε να τροφοδοτήσουμε την, ε, τις πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. Ε, να δούμε πώς φανταζόμαστε ότι θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα στο μέλλον. Θα πρέπει να το κάνουμε προκειμένου, όπως είπα, να τροφοδοτήσουμε τη διαδικασία λήψη λήψης πολιτικών αποφάσεων και η Στρατιωτική Επιτροπή θα δράσει σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, στηρίζοντας ε, τη διαδικασία ανάπτυξης των δυνατοτήτων. Φτάνω στα συμπεράσματά μου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου είχε ως στόχο να καταδείξει την βούληση των κρατών μελών να αναλάβουν από κοινού τι ευθύνε του σε θέματα ασφάλεια, σε θέματα άμυνα, Ξεκίνησε μια δυναμική και βρισκόμαστε στην αρχή μια καινούργια διαδικασία. Καθορίστηκαν χρονοδιαγράμματα και θα πρέπει να δουλέψουμε τους επόμενους μήνες και μέχρι τον Ιούνιο 2015, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στα 28 κράτη-μέλη με τους ε, αρχηγούς ΓΕΣ ε, εντός της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής θα εργαστούμε και εμείς με πολύ αποφασιστικότητα. Θα μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η Ευρώπη θα γίνει μάρτυρας πολλών συζητήσεων μεταξύ κομμάτων, ερετών εκπροσώπων, γενιών στα κράτη-μέλη. Εγώ από τη δική μου μεριά επιθυμώ μεταξύ άλλων θεμάτων που θα συζητηθούν να συζητηθούν και οι τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και γι' αυτό σας καλώ και εσείς να ε, τροφοδοτήσετε αυτές τις συζητήσει. Από την ε, θέση σε ισχύ τη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να γίνει ε, ένα παγκόσμιο παίκτη και να βαραίνει στην πύλη των κρίσεων ασφαλώς και πρέπει να κάνουμε ακόμα προσπάθειες αλλά η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και η απόφαση να ξεκινήσουμε μια καινούρια επιχείρηση στην, κεντρική, στην κεντροαφρικανική δημοκρατία ε, το αποδεικνύει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πτέραρχε για τις πολύ πλήρεις αυτές πληροφορίες που μας δώσατε. Δεν έχω να κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις Ενδεχομένω να πω κάτι, ενδεχομένως είναι και κάπω βέβαια νωρί για να το πούμε αυτό. Γενικά στις εργασίες σας λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη θεσμική συνεργασία και συνομιλία με το ΝΑΤΟ. Όσον αφορά το Αφγανιστάν, την περίοδο μετά το Αφγανιστάν, που θα ξεκινήσει ουσιαστικά στα τέλη του έτους και που ουσιαστικά θα απαιτήσει από τα περισσότερα κράτη-μέλη να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από το σημαντικότερο θέατρο επιχειρήσεων που είχαμε τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα του Αφγανιστάν μας απασχολεί ήδη πολύ και σας βέβαια στην Επιτροπή σας αλλά και τους εταίρους μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Θεωρείτε λοιπόν εσείς ότι ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στο Αφγανιστάν θα πρέπει ενδεχομένως να θέσουν σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα τα μέσα τους πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ε, ε, σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να κάνω στη συνέχεια κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, βλέπω ότι δεν αναφερθήκατε στην επιχείρηση Ουμπάμ στη Λιβύη. Στα πλαίσια ουσιαστικά των πέντε αποστολών κοινή εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας που λάβανε χώρα. Είναι λίγο περίεργο αυτό, δεν το αναφέρετε καθόλου. Δεν θα έπρεπε αυτό να αποτελεί τμήμα της παρουσίασής σας. Καταλαβαίνω ότι είναι μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο όμως θα έπρεπε να υπάρχει μια σημαντική στρατιωτική συνιστόσα και στις επιχειρήσεις αυτές. Τα καθήκοντα των επιχειρήσεων αυτών είναι σαφώς στρατιωτικά, ιδίως όσον αφορά την προστασία των θαλασσίων συνόρων. Εσείς στα πλαίσια της Στρατιωτικής Επιτροπής δεν ασχολείστε καθόλου αν μη τι άλλο με το συντονισμό των επιχειρήσεων αυτών μολονότι έχουν χαρακτηριστεί μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μία άλλη ερώτηση τώρα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, βλέπω ότι το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του ουσιαστικά μεταθέτει οποιαδήποτε απόφαση για τον Ιούνιο του 2014 εμείς πάντως περιμέναμε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, στο τελευταίο αυτό Συμβούλιο, θα καταφέρναμε τελικά να καταλήξουμε σε μία στρατηγική θαλασσίας ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε πάντως εσείς τώρα ότι υπάρχουν κάποια, αν μη τι άλλο, δείγματα διάρθρωσης κάπως της συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου αν μη τι άλλο να γνωρίζουμε ποιος κάνει τι και να καταφέρουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα συγκρούσεων αρμοδιοτήτων που έχουν προκύψει ιδίω στον τομέα της θαλασσίας ασφάλειας, να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνο για ποιο τομέα. Και κάτι ακόμα. Το θέμα των μη επανδρομένων εναρίων οχημάτων. Αναφερθήκατε προφανώς αυτό και είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια κάποια αυτονομία προς την χρήση των ε, οχημάτων αυτών. Θα μπορούσαμε κάπως να οριοθετήσουμε, μη τι άλλο όμως, τη χρήση τους, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χωρίς να θέτουμε απαραίτητα το ζήτημα αυτό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και χωρίς ουσιαστικά να λαμβάνουμε υπόψη ότι ε, οι Αμερικάνοι εταίροι μας χρησιμοποιούν πλέον τα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα με τρόπο θα έλεγα υπερβολικό πολλές φορές παραβιάζει και τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και το διεθνές δίκαιο. Ξέρετε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα του Targeted Killing ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σαφώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς μπορούμε εμείς τώρα να επιλύσουμε το πρόβλημα της χρησιμοποίησης των δικών μας μη επανδρομένων εναρίων οχημάτων όταν από την άλλη δίνουμε μια απόλυτη ελευθερία, συνδοσία θα έλεγα, στη χρήση των μη επανδρομένων αρίων οχημάτων από τους Αμερικάνους. Φοβάμαι ότι αυτό θα λειτουργήσει ως μπούμεραγκ τελικά κάποια στιγμή για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς να ασκήσουμε πίεση προκειμένου να τηρείται το διεθνές δίκαιο. Και ξέρετε ότι πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε αντίπεινα στην προσπάθειά μας να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο από τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ. Κατά την προετοιμασία λοιπόν της επόμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ θα έπρεπε να τεθεί και αυτό το ζήτημα. Και μια τελευταία παρατήρηση. Η αποστολή U4 στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Θα ήθελα να γνωρίζω προς αυτή και τη δική σας την άποψη. Το Συμβούλιο των Υπουργών αυτής της εβδομάδος έδωσε κάποιες διευκρινήσεις ως προς την αποστολή αυτή που εμένα κάπως με ανησυχούν ουσιαστικά τις βρίσκω κάπως αντιπαραγωγικές. Και ουσιαστικά Προσπαθώ εδώ πέρα να συγκρίνω την κατάσταση με την αποστολή στο Κονγκό το 2006. Ξέρετε ότι είχε γίνει μια ολόκληρη συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπήρχαν ορισμένοι ευρωβουλευτέ αλλά και κράτη-μέλη που θέλαν να περιορίσουν την αποστολή αυτή στην πρωτεύουσα μόνο τη χώρα και σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Βλέπω τώρα ότι την Δευτέρα οι υπουργοί αναφέρθηκαν στον Μπαγκή και σε μια χρονική περίοδο έξι μηνών. Είπανε έως 6 μήνες. Μα ξέραμε ούτως ή άλλως ότι η αποστολή αυτή αυτή τη στιγμή αρχίσει να αναπτύσσεται επί τόπου γιατί ξέρετε ότι ήδη από το Δεκέμβριο του 2012 μας λένε ότι υπάρχει μια απειλή γενοκτονίας, ήδη από το Μάρτιο του 2013 μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανθρωπιστικές μας ζητούν απεγνωσμένα να παρέμβουμε επί τόπου. προκειμένου να καταφέρουν και αυτές να επιτελέσουν το ανθρωπιστικό τους έργο. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο σας έλεγα. Πέρα από το πότε ακριβώς θα αναπτυχθεί τελικά η αποστολή αυτή, θα ήθελα και ως προς αυτό μια απάντηση, αλλά και κάτι ακόμα. Είναι σκόπιμο, είναι λογικό να έχουμε μια τέτοια αποστολή η οποία θα περιοριστεί μόνο στον μπανκί και μόνο για μια χρονική περίοδο έξι μηνών. Ξέρουμε βέβαια ότι εφόσον τελικά ε, αναπτυχθεί αποτελεσματικά η αποστολή αυτή, θα μπορούσε να την αλάβει στη συνέχεια και ο Οργανισμό των Εθνών. Αν γίνεται να απαντήσετε σε όλα αυτά, σα παρακαλώ πολύ. Δύο λόγια μόνο, κύριε Πρόεδρε. Αν υπάρχει μία αποστολή που πρέπει να την παρακολουθούμε ε, ήδη από την αρχή, είναι αυτή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Κονγκό παρακολουθήσαμε αυτό το σχεδιασμό και κάναμε και μια αξιολόγηση στο τέλος. Ε, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Το σημειώσαμε. Η κυρία Νικολάη, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Κύριε Πτέραρχε, θα σας θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, για την δημοκρατία την Αφρικανική Δημοκρατία χαιρετίζω την απόφαση να επέμβει εκεί, να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, βλέπω εδώ και τις συστάσεις που γίνονται και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η χρονική διάρκεια για την οποία μιλάμε εδώ. Και δεύτερο ερώτημα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να γίνουν εκεί ορισμένα πράγματα θα πρέπει να το δούμε και από οικονομική άποψη για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αν θέλετε την ασφάλεια ή τη συνεργασία. Έχουμε ανάγκη μιας ισχυρής ε, ε, αν θέλετε ε, ασφάλειας και βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πτέραρχε για την ε, για την ε, παρουσίασή σας η οποία ήταν αρκετά αισιόδοξη μετά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 12. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα ή σχέδια τα οποία θα εφαρμοστούν και θα, θα λειτουργούν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και κάτι τι άλλο από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισμένα και άρα περιορίζουν και τις στρατιωτικές δυνατότητες ή όχι υπάρχει μια παράγραφος που είναι ουσιαστικά δήλωση προαθέσεων τελείως θεωρητική και αφηρημένη για το τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη που πρέπει να διατηρήσουν την ασφάλεια και την ειρήνη. Ναι, αλλά πρακτικά πώς θα γίνει αυτό άμα συνεχίσουμε να έχουμε περιορισμό στις δυνατότητες μας και αυτό που είπε η κυρία Νικολάη για την πολιτική ασφάλεια στο κυβερνοχώρο έχει δίκιο. Λέγεται εδώ ότι το 14 θα οριστεί ένα πλαίσιο για το θέμα αυτό κατόπιν προτάσεως της ε, κυρίας Άστον. Πώς θα γίνει ακριβώς αυτό. Thank you, I would like to ask... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω για αυτή την ε, περίφημη Rapid Reaction Force, αυτές τις δυνάμεις άμεσης επέμβασης, ταχείας επέμβασης, γιατί ακούσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα εκεί και στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στο πώς λειτουργούν. Είπατε ότι θα ασχοληθείτε και με αυτό. Αλλά η πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο τι μορφή πήρε ε, για τις δυνάμεις αυτές θα ε, εξυγχρονιστούν κατά κάποιο τρόπο όλες οι χώρες που χρησιμοποιούν τις δυνάμεις αυτές δεν συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρήσεις της Ένωσης Ποια είναι σήμερα η σχέση μεταξύ των αντίστοιχων δυνάμεων του ΝΑΤΟ και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση για τα μη επανδρομένα αέρια οχήματα, για τα drones. Λοιπόν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από την έρευνα για τα οχήματα αυτά. Είναι γεγονός, αλλά αναφερθήκατε και σε δεοντολογικά και ηθικά προβλήματα που σχετίζονται με τα οχήματα αυτά. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο εντό των οποίων θα λειτουργούν τα οχήματα αυτά. Τι θα κάνετε σχετικά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Είπατε επίσης ότι θα προσπαθήσετε Παθήσετε να εντάξετε όλες αυτές τις συζητήσεις στην πολιτική διαδικασία. Πώς βλέπετε και εκεί ακριβώς τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ε, τρεις ακόμη ερωτήσεις θα ακούσουμε και μετά θα απαντήσετε. Ο κύριος Βανόρντεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Όχι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Απευθύνομαι στον τέραρχο Ντερουσιέ. Πάντως τα drones τελικά είναι το τελευταίο πράγμα που δαιμονοποιήθηκε από την αριστερά. Υπάρχει βαθύς αντιαμερικανισμός μεταξύ των αριστερών, της αριστεράς στο κοινοβούλιο που τελικά δεν αγαπούν αυτά τα drones και θα προτιμούσαν να γίνεται βομβαρδισμός γενικός ε, χωρίς στόχους παρά τα ε, να γίνεται στοχευμένο, ε, να γίνονται στοχευμένες επιχειρήσεις. Τώρα, για την... Για σας προσωπικά, τώρα που αναλάβατε την Προεδρία της Στρατιωτικής Επιτροπής ε, μετά από το ότι είσαστε εκπρόσωπος της Γαλλίας ε, στο ΝΑΤΟ κλπ. κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι λίγο γελίο τα ίδια άτομα να εμπλέκονται και από τις δύο όχθες αν θέλετε ε, δηλαδή δεν θα έπρεπε καλύτερα να έχει η Γαλλία ας πούμε δύο εκπροσώπους πώς αντιμετωπίζετε αυτό το διτό χαρακτήρα του λειτουργήματός σας έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία μόνο στρατιωτική επιτροπή η οποία θα εκπροσωπούσε ή θα εξυπηρετούσε αν θέλετε όλες τις δυτικές δημοκρατίες θα έλεγα εγώ στο δυτικό κόσμο αντί να έχουμε αυτό το διχασμό μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ρωτήσω και κάτι άλλο από την πείρα σας μπορείτε να μας πείτε πώς βλέπετε τις μελλοντικέ σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα ε, μεταγωγικά ε, ας πούμε ε, η σχέση μεταξύ των ναυτικών των δύο χωρών ποια νομίζετε ότι είναι ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα έλεγα ότι είσαστε ιδιαίτερα αισιόδοξο, ούτε απεσιόδοξο άλλωστε, αλλά θα ήθελα να πω ότι τα έγγραφά μας τα έγγραφα των ευρωπαϊκών ε, οργάνων είτε της, ε, των Υπουργικών Συνόδων είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα την πραγματικότητα που βιώνουμε στον κόσμο η οποία δεν είναι αισιόδοξη Υπάρχουν όλο και περισσότερες κρίσεις και καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι η μόνη ε, δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα είναι η στρατιωτική επέμβαση. Εδώ και δύο χρόνια μιλάμε για την κατάσταση στη Συρία. Χαίρομαι που προφανώς ε, κάποιοι στρατιωτικοί είναι αρκετά διστακτικοί όπως εσείς ενώ βλέπουμε να τους πολιτικούς να ενθουσιάζονται υπέρ της επιλογής στρατιωτικής ε, επέμβασης. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που δεν άκουσα από εσά κύριε Πτέραρχε ε, μιλήσατε για τις α, στρατιωτικές αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να εντάσσονται στο, σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά η πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί σωστά και για τις συγκεκριμένες αποφάσεις ουσιαστικά επικρατούν τα συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών. Θα Μακάρι να αναλάμβαναν οι πολιτικοί την ευθύνη πλήρως και μια από αυτές τις ευθύνες θα ήταν να καθίσουν να σκεφτούν το τι θα γίνει μελλοντικά όχι να δρούν εκ των υστέρων μόλις αναφιούν τα προβλήματα έχουμε άραγε εργαλεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη το σχεδιασμό μελλοντικών κινήσεων πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να παρέμβουμε εκ των προτέρων και διαμορφώσουμε μια κατάσταση αντί να παρέμβουμε εκ των υστέρων και για τα drones έχω μια άποψη διαφορετική από αυτή του κύριου Βαν Όρντεν Βέβαια δεν θα αναφερθώ σε αυτά στην προεκλογική μου εκστρατεία αλλά εμένα με με νοιάζουν οι ανθρώπινες ζωές ε, με ενοχλούν τα αθώα θύματα αυτών των μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων με ενοχλεί ότι χάνουν τις ζωές τους άνθρωποι που δεν ήταν στόχοι ουσιαστικά με άλλα λόγια η χρήση της πιο πρόσφατης τεχνολογίας θα πρέπει να βασίζεται σε ηθικές και δεοντολογικές αρχές αν θέλουμε αυτά τα οχήματα για αναγνώριση, ωραία, εντάξει, αλλά να τα χρησιμοποιούμε για να σκοτώσουμε αθώους συνανθρώπους μας, αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Πασκού, καλύτερη ερώτηση τελευταία φαντάζομαι. Um, I... Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες ιδέες που θα μπορούσαμε ίσως να τις σκεφτούμε. Θα ήθελα να αναφέρω όμως και δύο τεχνικά θέματα. Πρώτα πρώτα να πω ότι η Αυστραλία αναθεωρεί αυτή τη στιγμή τη θέση της για την αγορά αυτών των μη επανδρομένων αεροσκαφών για την παρακολούθηση των θαλασσών της. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεύτερο τεχνικό ζήτημα η κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία δεν απαιτεί ουσιαστικά βαριά πολιτική παρέμβαση αλλά κάτι το πιο ελαφρό, μια παρακολούθηση και εδώ θα πρέπει να δούμε τι συνδυασμό μπορούμε να εφαρμόσουμε δεν ξέρω η κατάσταση θα είναι σαν το μαλλί μπορεί να είναι ε, διαφορετική εν πάση περιπτώσει ξέρετε φαντάζομαι ότι ε, ε, θεωρούνται in the future and perhaps not all θεωρείται πιθανό να μπορεί να γίνει κάτι μέσω της χωροφυλακής κατά κάποιο τρόπο στην περιοχή ή κάποιες άλλες, κάποιων άλλων δυνάμεων ο, αντίστοιχων που θα μπορούσαν να φτιαχτούν στο μέλλον για την παρακολούθηση διαδηλώσεων ε, κτλ. Τώρα, το πολιτικό σκέλος, σκέλος παρακολουθώ αυτή τη στιγμή τι γίνεται στη Γερμανία ένας καινούριο ενθουσιασμός στη χώρα αυτή για να συμμετάσχει και πάλι σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υπάρχουν όμως πολιτικά θέματα ο Στάιν Μάιερ και άλλοι είπαν ότι θεωρούν ότι είναι έτοιμοι για να εκπαιδεύσουν το κοινό τι θα πει αυτό μέχρι τώρα οι, ε, οι ηγέτες μας προτιμούσαν να ήταν ουσιαστικά όμοιροι του κοινού και όχι εκπαιδευτές του, της κοινή γνώμης. Ας το σκεφτούμε λοιπόν πολύ καλά αυτό. Γιατί αν αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε τις κοινέ μας γνώμες και τους πολίτες μας ίσως καταφέρουμε να μειώσουμε τις αμυντικές δαπάνες αυτή μια ισορροπία μεταξύ των δύο θα ήταν ενδιαφέρουσα και σημαντική και επίσης θα πρέπει να αποδώσει μεγαλύτερη σημασία στο οικονομικό μέρος. Στο Αφγανιστάν έχουμε ένα κράτος που δεν ξέρουμε άμα αποσυρθούν οι δυνάμεις μας πώς θα λειτουργήσει και η οικονομία δεν έχει το κράτος αυτό θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα μετά την αποχώρηση από το Αφγανιστάν διότι μέχρι τώρα δεν ε, ε, κάναμε τίποτα για να δημιουργηθεί μια πραγματική οικονομία στο Αφγανιστάν. Το ίδιο ισχύει και για την κεντροαφρικανική δημοκρατία και την οικονομία της χώρας αυτής. Κάποιος όμως θα πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Και τέλος να πω ότι κάποια σχέση πρέπει να υπάρχει μεταξύ της περιφερειακής ανάπτυξης και της συλλογής πληροφοριών και να αρχίσουμε κάποια δουλειά σχετικά για να δούμε, για να βλέπουμε κάθε φορά αν χρειάζεται να παρέμβουμε και μετά την αποχώρησή μας, μετά την συγκεκριμένη επιχείρηση να έχουμε κάνει πολλά πράγματα ούτως ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία στη χώρα. Κύριε Πτέραρχη, έχετε ένα τέταρτο στη διάθεσή σας για να απαντήσετε σε αυτό τον εκτενή κατάλογο ερωτήσεων. Θα είμαι πολύ σύντομος. Απαντώντας με τη σειρά. Ε, διάλογος με τον ΝΑΤΟ μετά το Αφγανιστάν. Οι αρχηγοί ηγές ε, ε, πώς το σκέφτονται. Τι θα γίνει μετά το 2014 είναι το πρώτο ερώτημα. Τι δράση θα έχουμε στο Αφγανιστάν μετά το 2014. Η απάντηση τον Ιούλιο. Πριν τον Ιούλιο δεν θα ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι η εκπαίδευση. πώς θα εκπαιδεύσουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν όλα τα πολιτικά σενάρια. Δεδομένου ότι θα μειωθεί η παρουσία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ αρχίζουν σιγά σιγά να συζητούν το θέμα αυτό. Γιατί το θέμα έχει σχέση και με την εκπαίδευση της, ε, των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και με τις μάχημε μονάδε. Δεύτερο θέμα, στο οποίο σιωνιώνουμε πρόοδο, τη στιγμή που θα αναλάβει κάποια δέσμευση το ΝΑΤΟ, πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, διευκολύνει το ΝΑΤΟ και σε μη ζητήματα, σε μη καθαρά στρατιωτικά ζητήματα. Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά Πρέπει να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα. Πριν από κάποιο καιρό είχαμε τη συμφωνία Βερολίνο Plus. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια παρόμοια διαφορετική φύση συμφωνία για αυτό το ζήτημα. Τώρα, για το θέμα της ε, επιχείρησης Λιβύης. Από στρατιωτικής πλευράς η ε, δράση ήταν διμερής μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και της, ε, των ΗΠΑ ε, οι οποίες χώρες ε, εκπαιδεύουν τον μελλοντικό στρατό της Λιβύης. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, η ποιήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθαρά μη στρατιωτική. Η Στρατιωτική Επιτροπή δεν έχει καμία εμπλοκή. Σε ό,τι αφορά την στρατηγική θάλασσα, θα προβλέπετε ότι θα εγκριθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, συν, ε, από κοινού εργάζονται εντατικά και το επόμενο φθινόπωρο θα έχουμε στη Στρατιωτική Επιτροπή ένα προσχέδιο αυτής της στρατηγικής, θαλάσσιας στρατηγικής. Για τα μη επανδρομένα ε, οχήματα, το αφήνω στο τέλος, Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία πότε θα βρισκόμαστε επί τόπου. Ήδη βρισκόμαστε. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα. Ε, και έχει προχωρήσει στις πρώτες επαφές. Ο στρατηγός Πομπιές ε, έφτασε εκεί την περσμένη εβδομάδα στον Πάγκη για τις πρώτες επαφές με την Αφρικανική Ένωση, με τις ε, αρχές της Κεντρικής, Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και με την αποστολή της Γαλλίας που βρίσκεται επί τρόπου ήδη. Η διαδικασία ε, είναι, ε, ο σχεδιασ... αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται στο σχεδιασμό ε, ποιε δυνάμει, πόσε δυνάμει θα αναπτυχθούν και ε, πώ θα δράσουν. Αυτέ είναι πολύ σημαντικέ εργασίε που στο 90% των χωρών χρειάζεται να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν ξέρω πότε θα αναπτυχθεί η δύναμή μας. Το συντομότερο δυνατό είναι ο στόχος μας και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε γρήγορα προς όφελος της ασφάλειας. Και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια του Μαρτίου θα τα έχουμε καταφέρει. Οπότε έχουμε τον υπόλοιπο Φεβρουάριο και εκτός από το σχεδιασμό θα πρέπει να προετοιμάσουμε και την αύξηση των ε, δυνάμεών μας. Θα πρέπει στον πάγκι να κάνουμε τις κατάλληλες προετοιμασίες σε αποβουλάς υποδομής και υποδοχής. Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και πάλι να σας πω ότι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, σας το ανέφερα μόλις τώρα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ε, σχετίζονται με το γεγονό ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο ε, το θέμα και να κατανοούν με τον ίδιο τρόπο το πόσο επίγον είναι πέραν της ανθρωπιστικής διάστασης. Τώρα, τα, είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν στρατιωτικές δεσμεύσεις και να παρέμουν και με τη βία ε, ενδεχομένω ε, ανάμεσα σε φατρίες που αλληλοσφάζονται πολλές φορές. Παίρνει χρόνο για να καταλήξουμε σε κοινό όραμα. Ομοφωνία μεταξύ των 28 ε, ε, στα λόγια δεν είναι δύσκολη, είναι εύκολη. Α, αλλά από την, ε, ε, από την ανάληψη των δεσμεύσεων, μην ξεχνάμε, ε, από την και μετά, θα έχουμε και άλλα γεγονότα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση. Οπότε δεν ξέρω σε έξι μήνες, τον Οκτώβριο, πούμε, αν θα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Όμως, τα κράτη-μέλη θέλουν όλα να είναι στη θέση τους έτσι ώστε να κάνουμε τη διαφορά έτσι ώστε η Αφρικανική Ένωση σε μερικούς μήνες να πάρει τη σκητάλη. Οπότε έχουμε δύο ε, άξονες δράσης. Πρώτον, ε, να καταστήσουμε την ασφάλεια και την ειρήνη στον πάνκι. ασφαλώς περιοριζόμαστε στον Πάγκη, αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ε, θα πρέπει οι στόχοι μας να, είναι, ε, να συνάδουν με τις ε, δεσμεύσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα μέσα που θέτουν στη διάθεση της κοινή δύναμης. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας ε, θα θέσουμε σε λειτουργία ε, ε, μέσα προστασίας εναντί επιθέσεων στον κυβερνοχώρο συμπεριλαμβανομένων και του Μπάνκι και, της, και του στρατιού της Λάρισας. Εκεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα ε, συνεργάζεται με το κέντρο αριστεία του Τάλιν στην Εστονία. Και ε, δεύτερον, στην Στρατιωτική Επιτροπή έχουμε επεξεργαστεί ένα έγγραφο στρατηγική ε, για την ασφάλεια την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Αλλά οι δράσεις δεν είναι στρατιωτικές δράσεις, κοινές στρατιωτικές δράσεις, θα είναι δράσεις από τα κράτη-μέλη. Τώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η συνεργασία, είναι πολύ περίπλοκο. Πολλοί το προσπάθησαν, αλλά αντιμετώπισαν δυσκολίες. Όταν έχουμε ε, ε, αν, όταν έχουμε με έξι μήνες διαφορά δύο συναντήσεις κρατών, αρχηγών κρατών κυβερνήσεων ε, και πριν από την πρώτη από αυτές ε, οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων λένε ότι θα πρέπει να σφίξουμε τη σχέση με τον ΝΑΤΟ αλλά δεν το κάνουμε. Προειδοποίησα τον πρώτο της, ε, της Επιτροπής του ΝΑΤΟ που θα έρθει νομίζω το απόγευμα εδώ να σας μιλήσει. Τον προειδοποίησα για το τι θα κάνουμε στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Αλλά η δική μου επιτροπή, αλλά ε, που δεν είναι, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στο κέρας Αφρικής ε, με τις δύο αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν θα λύσουμε τα προβλήματα μέσω της ενοποίησης των στρατιωτικών επιτροπών. Όχι πρέπει να συνεργαστούμε. Η συνεργασία μας, παρόλο που δημοσίως λέω ότι λειτουργεί, δεν λειτουργεί όσο θα έπρεπε. Σταδιακά λοιπόν θα γίνουν ε, οι αλλαγές. Ε, για πολιτικούς λόγους δεν μπορούμε να πάμε πολύ γρήγορα. Ατύπως όμως κάνουμε πρόοδο στη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών. Με, για τους μειωμένους ε, αμυντικού προπολογισμού, ναι, όλοι μα λειτουργούμε με μειωμένου προπολογισμού. Οι αρχηγοί ΓΕΣ, ε, οι αρχηγοί, ε, συγγνώμη, εξετάζουν διάφορες αναλυτικές λύσει. για το πώ μπορούν να κάνουμε τα ίδια πράγματα με λιγότερους πόρους. Οι τα περιφερειακά κλάστερ συνεργασίας, για παράδειγμα στη Βαλτική, στι χώρε του Βόρα, η B4, ε, είναι πρωτοβουλίε που επιτρέπουν αύξηση των συνεργειών μεταξύ των κρατών μελών. Με αυτό το στόχο. Στην εκπαίδευση, για παράδειγμα. Αυτό που κάνουν οι χώρε τη Βαλτικής, το, η Πολεμική Ακαδημία της Βαλτικής, ε, είναι πρωτοβουλίε οι οποίε θα αντιγραφούν και αλλού αυτό δεν σημαίνει δημιουργία μιας πολεμικής σχολής ή ενός ευρωπαϊκού κολεγίου, ε, ε, ε μιας ευρωπαϊκής πολεμικής ακαδημίας. Όχι. Ε, είναι περιφερειακές μονάδες ως αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ ενός αριθμού κρατών μελών. Ταχεία αντίδραση. Σύνος κορυφής εξέφρασε την επιθυμία της να ασχοληθούμε με το θέμα της ταχείας αντίδρασης. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τις ε, μάχημες μονάδες που είναι εξαιρετικό ε, ε, εργαλείο. Και το ΝΑΤΟ έχει την, τη δύναμη αντίδρασης, δύναμη ταχείας αντίδρασης. Είναι πολύ σημαντικά μέσα εργαλεία που έχουμε. Μέσω της ε, του πολυεθνικού χαρακτήρα των μάχημων μονάδων μας 1.500-2.000 ε, ε, ανδρών δημιουργούνται συνεργίες, συνέργειες αλλά είναι μικρές αυτές οι μονάδες δεν μπορούν ασφαλώς να αναλάβουν όλο το μπάγκι στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αλλά μπορούν να αναλάβουν για παράδειγμα το αεροδρόμιο του μπάνκι. οπότε δεν είναι μόνο το, το πλεονέκτημά τους δεν είναι ε, ότι είναι υψηλές δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες, αλλά οι μάχημες μονάδες μας έχουν το χαρακτηριστικό ότι ε, είναι πολυεθνικές. Δημιουργούν συνέργειες. Θα πρέπει να σκεφτούμε όμως τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των στερεωτικών σωμάτων στις χώρες στις οποίες αναπτυσσόμαστε. Θα πρέπει δηλαδή να αναζητήσουμε ένα καινούριο εργαλείο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να απαντούμε ταχύτατα σε περιπτώσεις κρίσεων. Οι μάχημες μονάδες θα υποστηρίζουν απλώς ε, τις υπόλοιπες δράσεις. Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει θα είναι μια δομή πολύ διαφορετική από τις μάχημες μονάδες, αλλά και πολύ διαφορετική από τη μονάδα ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Θέσατε ένα άλλο ερώτημα όσον αφορά τα αεροπλανοφόρα και την χρήση τους από την uh, Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ δεν εκπροσωπώ τη Γαλλία, επομένως δεν μπορώ να μιλήσω για τη χώρα αυτή. Ελπίζω πάντως ότι στο μέλλον θα καταφέρουμε συλλογικά να αποφασίσουμε για το πώς θα συνεργαστούμε με το 2020, το 2030, όχι μόνο η Γαλλία και η Αγγλία, αλλά και η Ιταλία, η Ισπανία, πώς θα καταφέρουμε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε μη συμβατικά αεροσκάφη, τα οποία θα είναι σε θέση να κάνουν πτήσεις αναγνώρισης, να κάνουν επιθέσεις, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, όχι μόνο στα πλαίσια της UCAV, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες συλλογικές τέτοιες ε, μονάδες. Να περάσω τώρα στο ερώτημα των μη επαντρωμένων ε, ενέργειων οχημάτων. Ουσιαστικά έχουμε ένα μια στρατιωτική μονάδα η οποία αυτή είναι πάρα πολύ καλύτερη ουσιαστικά. Το θέμα είναι ότι όταν εκτοξεύδουμε ένα πύραυλο για παράδειγμα δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Μετά από τρία λεπτά απλώς θα καταστρέψει μια περιοχή. Όταν χρησιμοποιείτε ένα μη επανδρομένο ενέργειο όχημα έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Ανα πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε την πορεία του. Εγώ υπήρξα πιλότος της πολεμικής αεροπορίας σε πτήσεις αναγνώρισης βγάζαμε τη δική μου την εποχή απλώ κάποιε φωτογραφίε. Τώρα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε πραγματικά βίντεο. Γνωρίζουμε ακριβώ την παραμικρή κίνηση. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου πώ ακριβώ κινείται, από πότε βγαίνει από το κτίριο, πότε μπαίνει στο κτίριο του Κοινοβουλίου. Με έναν ύποπτο ακριβώ το ίδιο πράγμα. Μπορούμε να συλλάβουμε, αν θέλετε, κάποιον, όχι απαραίτητα να τον σκοτώσουμε. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζετε ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και δεν αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στα drones που χρησιμοποιεί η CIA ή άλλοι φορείς. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα πραγματικά σώζουν ζωές. Στο, Αφγανιστάν, στο Αφγανιστάν έχουν σώσει τις ζωές των στρατιωτών μας. Ακριβώς επειδή είχαν εντοπίσει ότι υπήρχαν κάποιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των δικών μας των στρατιωτών. Με τη χρησιμοποίηση όμως αυτών των μη επανδρομένων ενέργων οχημάτων καταφέραμε να καταστρέψουμε ε, σε εκρηκτικούς αυτούς μηχανισμούς. Τα δικά μου τεγόνια βέβαια δεν θα έχουν τις ε, ίδιες ευκαιρίες με μένα να γίνουν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, ακριβώς επειδή στο μέλλον θα έχουμε πάρα πολλά αεροσκάφη αναγνώρισης, τα οποία τελικά θα είναι τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα. Πρέπει λοιπόν να δούμε εμεί πώς συλλογικά θα διαχειριστούμε αυτές τις νέες ευκαιρίες που προβάλλουν μπροστά μας και όντως τίθενται αυτά τα ηθικά διοντολογικά ζητήματα. Εμείς θα χειριστούμε τα συστήματα αυτά με βάση την Ευρώπη στα πλαίσια μιας κοινοτική ε, αποστολής ή θέλουμε να είμαστε πραγματικά παρόντες στη χώρα που αναπτύσσονται τα νέα αυτά μέσα. Αυτό σαφώς θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και αυτή η συζήτηση θα πρέπει να λάβει χώρα σε πολιτικό επίπεδο και θα πρέπει βέβαια να εμπλουτιστεί, να τροφοδοτηθεί και από τη δική μας την εμπειρογνωμοσύνη, με απότερο στόχο ίσως κάποια στιγμή να αποφασίσουμε σε πολιτικό επίπεδο ότι πρέπει να έχουμε πλέον ένα νομικό πλαίσιο, κάποιες νομικές διατάξεις σε σχέση με τη χρήση των αυτοματοποιημένων αυτών συστημάτων. Αυτός όμως είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμεθα πλέον. Θα υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες τέτοια εναέρια οχήματα μη επανδρομένα στο μέλλον. Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα, πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό και ουσιαστικά ακολουθεί την όλη πορεία που ξεκίνησε από την ανακάλυψη των αεροσκαφών. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια τεχνολογική επανάσταση η οποία επηρεάζει όχι μόνο το στρατοτικό τομέα αλλά και την καθημερινή μας ζωή. Και από αυτού επίσης να πω ότι Όσον αφορά την θαλάσσια αποπτία, ήδη πάλι έχουμε ένα καταπληκτικό μέσο το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Πώς όμως θα καταφέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε, με ποιο τρόπο. Εγώ ελπίζω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον έχουμε ένα τόχερον 2 δηλαδή τη χρησιμοποίηση δορυφόρων προκειμένου να καταφέρουμε να εντείνουμε όλες αυτές τις αποστολές εποπτείας, παρακολούθησης, ελέγχου των θαλασσίων μεταφορών και θαλασσίων κινήσεων και θα μπορούσε αυτό το σύστημα να συνδεθεί και με τη χρησιμοποίηση των μη επανδρομένων εναρίων οχημάτων που συστούσαμε πριν από λίγο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό και ποιοι είναι οι διάφοροι φορεί που θα χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό, προκειμένου τελικά να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια αρνητικά φαινόμενα όπω οι παράνομε διακινήσει, η παράνομη μετανάστευση κ.ο.κ. Ουσιαστικά μέσω των νέων αυτών συστημάτων πρέπει από κοινού να καταφέρουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, μια κοινή ανάλυση των δυνατοτήτων που μας δίνονται από τα νέα αυτά μέσα. Πρόεδρος, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αναφερθήκατε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στο πώς μπορούμε μάλλον να ενημερώσουμε καλύτερα το κοινό. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα σε σχέση με αυτό. Κάτι πάρα πολύ εύκολο, το οποίο ήδη κάνω εγώ. Όσον αφορά τους νέους στρατιωτικούς, προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι για έναν πολίτη ή για έναν αξιωματικό, για παράδειγμα, στην Κύπρο, στη Φιλανδία, σε κάποια χώρα της Βαλτικής, η άμυνα και η ασφάλεια δεν έχει την ίδια έννοια που έχει στην Πορτογαλία, τη Γαλλία ή κάποιες άλλες χώρες. Προσπαθούμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τους νέους αυτούς στρατιωτικούς ως προς τις υφιστάμενες προκλήσεις κάθε φορά με βάση τη γεωγραφική ζώνη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε το Δεκέμβριο ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2015 η ύπατη εκπρόσωπος θα πρέπει να υποβάλει μία αξιολόγηση των προκλήσεων ασφάλειας και πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν. Εγώ ελπίζω ότι η όλη διαδικασία που θα οδηγήσει στην αξιολόγηση αυτή θα είναι μία ανοιχτή, διαλλακτική διαδικασία όπου θα μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, στρατιωτικοί και μη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς και ότι θα μπορέσουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικά να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουμε συλλογικά όλοι μας. Πρόεδρος, κύριε Πτέραρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ, κάνετε την παρουσίαση και απαντήσατε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ξέρετε ότι και στα πλαίσια των διαφόρων οδικών χαρτών που έχουμε είναι και αυτό ότι τους επόμενους μήνες θα πρέπει να έχουμε μία αξιολόγηση. Μολονότι βέβαια σε 1,5 χρόνο, αν θέλετε, έχουμε αυτή τη σύνοδο ορόσημο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία θα πρέπει, ενδιάμεσα, τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευχαρίστηση να σας ξαναδούμε μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Ωστόσο, για όσους θα έχουν την τιμή να συμμετέχουν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξέρετε ότι θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας ξαναδούμε εδώ σε αυτό το θεσμικό όργανο. Κύριε Πτέρερχε, σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Όπως είπε και η Άννα Γκόμες, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η νέα αυτή επιχείρηση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο την τύχη ήδη από την αρχή της αποστολής αυτής να μπορούμε να ασκούμε εμεί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πίεση για περισσότερες πληροφορίες και μια πιο πλήρη ενημέρωση για την αποστολή αυτή, εμένα να σας πω μου έκανε πραγματικά εντύπωση η διαφορά ανάμεσα σε κάποιες πολιτικές δηλώσεις που γίνανε από ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία δεν καταλαβαίνω που τάχθηκαν υπέρ ή κατά της ε, επιχείρησης αυτής, Πρέπει να σας πω ότι ορισμένοι κάναν όμως κάποιες ιδιαίτερα περιπετειώδεις θα έλεγα δηλώσεις και παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι ε, η επιχείρηση αυτή με το εύρος της, με την ταχύτητά της ε, απέχει πολύ από αυτό το οποίο είχαν ανακοινώσει ορισμένοι και από αυτό το οποίο φοβόντουσαν κάποιοι άλλοι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στο μέλλον μια πιο ακριβή αξιολόγηση όσον αφορά αυτήν και τις μελλοντικές αποστολές. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πτέραρχε και τώρα να καλωσορίσουμε την κυρία Αρνού η οποία έχει φτάσει. Συνάδελφοι, έχουμε κάπως αργήσει. Δεν θα κάνω μια μεγάλη εισαγωγή. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην κυρία Αρνού. Ε, γιατί τελικά η Αζάνς πρέπει να είναι το πιο ευχαριστημένο κοινοτικό όργανο σχετικά με το τι έχει να κάνει πάρα πολλές εντολές ανα, σας ανατέθηκαν η τροφοδοσία η εναέρια η επικοινωνία μέσω δορυφόρων η ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή ε, τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που κουβεντιάζαμε πιο πριν ε, έχετε πάρα πολλή δουλειά να κάνετε και υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο επί μακρόν έχουμε συζητήσει με άλλες επιτροπές ε, και αυτό είναι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που ζητήθηκαν για την έρευνα που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα βεβαίως από οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι η ο οργανισμός σας, ε, η agency αυτή που εκπροσωπείται πραγματικά έχει πολλά πράγματα να κάνει ε, αυξάνει με μια έννοια αν θέλετε την αναγνωρισιμότητά της ή την ορατότητά της στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα ε, αλλά εν πάση περιπτώσει καλύτερα να σας δώσω το λόγο ε, για να μας δώσετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες όμως ε, να σας πω ότι εμείς οι περισσότεροι από εμά ε, από την πολιτική σκοπιά θεωρούμε ότι δεν ήταν αρκετά φιλόδοξα αυτά που σας ανατέθηκαν θα μπορούσαν να είχαν ανατεθεί κι άλλα λοιπόν έχουμε μια ωρίτσα στη διάθεσή μας ελπίζω να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά έχετε το λόγο κυρία μου euh, ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα για να συζητήσω τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από ό,τι κατάλαβα έχετε ήδη συζητήσει τα συμπεράσματα αυτά, τα συζητήσατε το στρατιωτικό σκέλος με τον τέραρχο προηγουμένως και άλλες, άλλα σκέλη με άλλους υπεύθυνους. Για μας τα συμπεράσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί πραγματικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας ανέθεσε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Εγώ ήδη εξ αρχής ήμουν πεπισμένη ότι θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία αυτή για να μπορέσουμε να προωθήσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα βέβαια, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα όπως είπα, προγράμματα αφενός ή να δούμε τι κίνητρα και πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για συνεργασίες και συντονισμό. Ε, μέχρι τώρα το ότι οι προτεραιότητες δίνονται σε στρατιωτικά θέματα δεν ήταν κάτι το προφανές. Τώρα όμως βλέπουμε να θεωρείται προτεραιότητα ε, αυτό το στρατιωτικό σκέλος και στρατιωτικές δράσεις. Βεβαίως όλα αυτά περνάνε από μια συνεργασία, συντονισμό, συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένη εντολή και αυξημένα κίνητρα στα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν. Ε, φαντάζομαι ότι το έχετε ήδη ξανακούσει από άλλους ότι ε, ε, τα κράτη-μέλη που δεν αποφάσισαν ομόφωνα ορισμένα πράγματα ε, σημαίνει ότι κάθισαν και το σκέφτηκαν πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Τελικά όμως μας έδωσαν μια εντολή από τους, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Σκέφτηκαν πολύ, μας ε, διαμόρφωσαν την εντολή αυτή και τώρα έχουμε αυτή την εντολή. Πρέπει να υπάρχουν πραγματικά προγράμματα, σημαντικά προγράμματα, αναφέρατε μερικά αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη ε, την ε, τροφοδοσία την αναέδεια την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κλπ. Νομίζω ότι ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί καταλήξαμε σε αυτό το, συμπέρασμα διότι όλοι μας συλλογικά η βιομηχανία, τα κράτη-μέλη, ε, οι κοινωτικές υπηρεσίες ε, όλοι συγκλίναμε προς τον ίδιο στόχο και έτσι ε, καταλήξαμε στο να δίνεται προτεραιότητα σε στρατιωτικές ενέργειες που περνάνε όμως βεβαίως από την συνεργασία και το συντονισμό. Αυτό ήταν ο ρόλος του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού, αυτό ήταν αυτό που τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπα ότι εκπρόσωπος και ε, άκουσα αυτά που είπε και ο πρόεδρος ο προηγούμενα στον Τέραρχο Ρουζιέ για το ότι η πιθανότητα δεν θα είναι η τελευταία αυτή η συνεδρία, η συνεδρία στην οποία παρευρισκόμεθα εδώ. Ελπίζω και εγώ να ξαναέρθω εδώ να σας ενημερώσω. Γιατί αποδίδουν μεγάλη σημασία η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο ε, και αυτά συμμετέχουν και συγκλίνουν εμπολείς και τα εθνικά κοινοβούλια φαντάζομαι με τα οποία έχετε ήδη συζητήσει ε, μπορούν να συμμετάσχουν. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια δυναμική μέσω όλων αυτών των φορέων που συζήτησαν και βεβαίω σημαντικό ρόλο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε έπαιξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εκτός των άλλων ήταν και ιδιαίτερα ρεαλιστική στην προσέγγισή της. Πολλοί από εσά ή από εμά βρεθήκαμε στο Μόναχο γιατί, πριν από δέκα μέρες για τη συνδιάσκεψη για την ασφάλεια και εκεί είδαμε ότι ακριβώς τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η παρουσία όλων μας και τα λοιπά επηρέασαν την ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων για την ε, συνεργασία, για το συντονισμό και είδαμε ότι η Γερμανία ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις αν θέλετε για να ε, αναλάβει ε, δράση για ενάντια στην κρίση, σε διάφορες κρίσεις κτλ. Τώρα, ε, να δούμε πιο συγκεκριμένα τι έχουμε να κάνουμε εμείς σαν ε, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Άμυνα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα άλλα κοινοτικά όργανα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα να διατηρήσουμε τη δυναμική τώρα για τα επιμέρους προγράμματα ε, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, θα απαντήσω ρωτήσεις αν υπάρχουν βεβαίως, αλλά δεν έχουμε ε, πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ο αναέριος, ε, αναέ, ε, ο ανεφοδιασμός, όπως είπατε, έχει υψηλή προτεραιότητα, την οποία ευλόγησαν οι διάφορες κυβερνήσεις. Ε, η, η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ασχολήθηκε με το θέμα αυτό για το ειδικό, ειδική, ε, ειδικό ανεφοδιασμό συγκεκριμένων τύπων στρατιωτικών αεροπλάνων. Η Ολλανδία επίσης ασχολήθηκε με το, με το θέμα αυτό και, και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε όλο και περισσότερο συνέργειες με τους στόλους αν θέλετε ε, των, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ. Τώρα, για τα μη επανδρομένα αέρια οχήματα, για τα drones, φαίνεται αυτό, ότι αυτό είναι το κατεξοχήν θέμα συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και ε, ε, Βεβαίως υπάρχουν τέτοιου είδους οχήματα παρατήρησης που τα ανέφερε και ο Κιουπτέραχος του Ρουζιέ θα πρέπει να ε, υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η Κομισιόν και θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κανονιστικές αυτές διατάξεις και να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε τη νέα τεχνολογία θα πρέπει να δούμε, να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά ε, ευρωπαϊκών drones για παρατήρηση και θα πρέπει να δούμε ε, τι αγοράζουν αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη, ε, τι υλικό σκέφτονται ότι πρέπει να αγοράσουν και βεβαίως υπάρχουν και τα πολύ σοβαρά θέματα της πιστοποίηση της μελλοντικής γενιάς τέτοιων μη επαδρομένων αέριων οχημάτων. Αυτά τα θέματα είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί υπάρχει μια πρόσθετη, μια ε, προσθέμενη αξία σε τέτοιου είδους θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά ε, υπάρχει το δορυφορικό κέντρο επίσης το οποίο ανέφερε ο πτέραρχος προηγούμενα ε, τέτοιου είδους κέντρα και δράσεις ε, που σχετίζονται και με στρατιωτικά και με πολιτικά θέματα, στρατιωτικά και μη στρατιωτικά, θέματα σαν και αυτό το κέντρο είναι πολύ σημαντικά. Από εκεί και πέρα για την ασφάλεια στον κυβέρνο χώρο θα είμαι ειλικρινής. Δεν έχουμε πο, κάνει πάρα πολλά πράγματα εδώ. Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι συγκλονιστικές. Θα πρέπει να φροντίσουμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε τα στρατηγία μας, τα γενικά επιτελεία ή και τους ιδιώτες. Εν πάση περιπτώσει το καλύτερο ε, το καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσετε ε, θέματα για τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ και ε, γι' αυτό δεν θα επιμείνω εγώ. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με τον ΝΑΤΟ. Ε, κάτι τι άλλο που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα συζητηθεί με το, από τους Υπουργούς Άμυνας στην επόμενη σύνοδό τους είναι η ασφάλεια των θαλασσών. Εμείς θα υποβάλουμε προτάσεις συμπληρωματικές προς μια γενική στρατηγική που φαίνεται να διαγράφεται αυτή τη στιγμή και ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τώρα, από εκεί και πέρα να πω βέβαια ότι οι εντολές που πήραμε είναι πραγματικές προκλήσεις για μας πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτούς που ε, έχουν ειδική και γνώσεις και σε οικονομικό και σε χρηματοπιστωτικό δημοσιονομικό επίπεδο για να δούμε τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει σε μονομερές ή ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί παίζει ρόλο βεβαίως στο οικονομικό μέρος οι δικές μας οι δομές είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν πάρα πολύ εύκολα τη συνεργασία. Μιλάμε δηλαδή για εθνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι σαφώς εθνικές, κυρίαρχες εθνικές και δεν είναι φτιαγμένες απαραίτητα για να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως ίσως θα πρέπει να δούμε το οικονομικό μέρος και να δούμε ότι ε, ε, ε, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα γιατί, γιατί τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα ούτε από οικονομική άποψη αν θέλετε ε, την ίδια στιγμή να ξεκινήσουν ε, κάποιες ε, δράσεις, κάποιες προσπάθειες, κάποιες επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι θα εναρμονίσουμε τα χρονοδιαγράμματα που ακολουθούν τα κράτη-μέλη αλλά θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μια και ένα κοινό σχεδιασμό, μια, ένα να μπορέσουμε να οργανώσουμε και την οικονομική στήριξη κάποιων δράσεων από κοινού για να μπορέσουν να γίνουν πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την Κομισιόν, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε κάποια κίνητρα στα κράτη-μέλη να δρουν από κοινού και σύγχρονα αν θέλετε. Τώρα, για κάποια από τα θέματα που μας ανατέθηκαν, το μας είπαν να αρχίσουμε ήδη από το 14 και για άλλα από το 15. Θα προσπαθήσουμε να δράσουμε λοιπόν α, ήδη αν μπορούμε από το τέλος του εξαμήνου, του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς. Τώρα... Θα πρέπει να δούμε και το θέμα της επικάλυψης, της διπλής χρήσης αν θέλετε. Μίλησα για τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, ε, νέες τεχνολογίες, κάποια, ως, κάποια ε, εργαλεία που έχουν διτή χρήση. Αυτά όλα είναι ε, η πρώτη υποψήφια αν θέλετε για να αναλυφθεί η επεξεργασία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άρα για να δοθούν και επιπλέον κονδύλια ε, γιατί, διότι η διτή χρήση σημαίνει ότι υπάρχει και στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση και άρα ίσως είμαστε πιο ελεύθεροι να δράσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο πρόεδρος μίλησε για την προπαρασκευαστική δράση. Αυτό έχει αρχίσει να μας απασχολεί. Μιλάμε με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου η προπαρασκευαστική αυτή φάση να τροφοδοτηθεί με συγκεκριμένες δράσεις για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Θέλουμε και τους στόχους της πολιτικής αυτής να καλύψουμε, αλλά και τις νέες δράσεις, τις τεχνολογικές που έχουμε ξεκινήσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο στόχος μας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι ο ακόλουθος. Να είμαστε έτοιμοι για την περίοδο 2016-2018 έτσι ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε και μία αξιολόγηση της προπαρασκευαστικής αυτής δράσης για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Ο δικός σας ο ρόλος επ' αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εν κατακλείδη και για να αφήσω και χρόνο έπειτα για τις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να πω ότι ε, δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή κάποια ραγδαία θεσμική αλλαγή. Δεν τροποποίησαμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, όπως το είπατε και εσείς Πρόεδρε, δόθηκαν απλώς σημαντικά καθήκοντα σε αυτόν τον οργανισμό που συνάδουν όμως με την αποστολή του όπως προβλέπεται από τη συνθήκη και όπως το είπατε κύριε Πρόεδρε Πιστεύω ότι ουσιαστικές τροποποιήσεις θα δούμε με βάση την αντίδραση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων στις προτάσεις που εμείς θα καταθέσουμε για τα προγράμματα, τα συμπληρωματικά προγράμματα τα οποία θα προτείνουμε, ιδίως στον τομέα της θαλάσσης ασφάλειας και όσον αφορά αυτά τα φορολογικά κίνητρα. Μία τελευταία παρατήρηση και ενδεχομένω κάπως προσωπική με την αδειά σας κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πραγματικό άλμα όσον αφορά τη δέσμευση των κρατών μελών για τις κοινέ δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν οι Υπουργοί Άμυνας πραγματικά αρχίσουν να αισθάνονται άνετα στο ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο. Νομίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας είναι αν θέλετε ο κατάλληλος χώρος για τη συνεργασία αυτή και ξέρετε είναι το τελευταίο σκέλος αν θέλετε της οικογένειας το οποίο δεν είναι ακόμα εντελώς ενταγμένο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα δούμε μια ειλικρινή δέσμευση των κρατών μελών σε θέματα άμυνας και σε θέματα στρατιωτικών δυνατοτήτων όταν πραγματικά ενταχθούν οι Υπουργοί Άμυνα σε αυτό το πλαίσιο και τότε θα μπορούμε να πάρουμε και συγκεκριμένε αποφάσει όσον αφορά του αμυντικού προπολογισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουν και οι Υπουργοί Άμυνα να συνεδριάζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ω ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα αναδιοργανώσαμε κάπω τη διάρθρωσή μα ε, έτσι ώστε να έχουμε μία διεύθυνση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα η οποία να έχει ως αποστολή να συνεργάζεται με τα διάφορα θεσμικά όργανα, τους διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια αρχική φάση. Έχουμε τροποποιήσει απλώς το οργανόγραμμα. Αυτό που όμως θέλουμε είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας να μπορεί να συνεργάζεται όλο και περισσότερο με τα Εθνικά Υπουργεία Άμυνας προκειμένου αυτά με τη σειρά τους να ενταχθούν περισσότερο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, να μπορέσουν να συνδιαλλαγούν με άλλους φορείς και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να αναπτύξουμε περισσότερο τόσο τις δυνατότητες που είναι ο δικός μου τομέας, αλλά και μια γενικότερη νέα νοοτροπία για τον τομέα της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, με πολλή ικανοποίηση ακούσαμε το τελευταίο σας σχόλιο, γιατί η εμπλοκή, η δέσμευση των Υπουργών Άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντική. Ο κ. Φανόρντεν ε, λείπει, ε, ναι το είπα και εγώ ότι είναι κρίμα. Ήθελα πολύ και εγώ να ανταλλάξω απόψη μαζί του. Ξέρω ότι θα του είχατε απαντήσει, οπότε μπορώ να το τα περάσω. Τώρα, ε, ο ρόλος της άμυνας ε, σίγουρα μπορεί να είναι πολύ σημαντικός στην, στον εξευρωπαϊσμό ε, των, των συναντήσεων των Υπουργών το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, υπηρεσία σας ε, λαμβάνει χώρα στο περιθώριο των ε, συναντήσεων των Υπουργών Άμυνα και ξέρω ότι στις δικές σας συναντήσεις ενδεχομένως είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή. υπάρχουν, τα δικά σας θέματα άπτονται άμεσα των οικονομικών ζητημάτων, οπότε αυτό με οδηγεί στην δική μου ερώτηση. Ε, λάβατε κάποιες εντολές από το, από το, από τη σύνολο Κορυφής. Θα ήθελα να σας ε, πω αν συζητήθηκε καθόλου ο προπολογισμό σας, γιατί ο προπολογισμό σας έχει μείνει στάσιμος τα τελευταία χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι ε, εξασφαλίσατε την αναγνώρισή σας, σας ανέθεσαν πολλά πράγματα, τον οδικό χάρτη και άλλα. Αλλά πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να βάλουν και το χέρι στην τσέπη. συζητήθηκε κάτι τέτοιο. Από τα σχόλια κάποιων συναδέλφων ε, από την άλλη μεριά της ε, μάχης ε, αντελήφθη ότι μάλλον δεν συζητήθηκε. Τέσσερις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο αντιπρόσωπος Παλέτσκι καταρχήν έχει το λόγο. Thank you for your comprehensive and clear statement. Κύριος Παλέτσκης, ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη δυνατότητα συνεργασίας ή την πραγματική συνεργασία που λαμβάνει η χώρα ανάμεσα στην υπηρεσία σας και τις συνδεδεμένες ε, χώρες, συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες. Ε, με τις χώρες, για παράδειγμα, της ανατολικής εταιρικής σχέσης, όπως η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ουκρανία. Έχετε επαφές, συνεργασία, σχέδια με αυτές τις χώρες. Και αν ναι, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία. Ευχαριστώ, κύριο Πάσκου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ε, εγώ φαντάζομαι τις μέρες που ε, θα είναι και οι Υπουργοί Οικονομικών παρόντες ε, στις συναντήσεις του ε, Διοικητικού Συμβουλίου σας. Γιατί είναι πολύ σημαντικοί αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε θεωρείτε ότι το, Συμβουλίο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε τη στροφή που όλοι περιμέναμε σε θέματα άμυνας. Ε, προφανώς το συμπέρασμα είναι ε, ότι η άμυνα είναι σημαντική αλλά χωρίς ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Ε, δεύτερον, σκέφτεστε τη χρήση των μη επανδρομένων οχημάτων σε σχέση με την πολιτική θαλάσσιας ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρόμπερκ. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίασή σας. Σε ό,τι αφορά κορυφής θα ήθελα να ρωτήσω το εξής ακούστηκε η ιδέα της συνένωσης και διαμοιρασμού του pooling and sharing της συνένωσης και κοινή χρήσης των μέσων Ξέρω ότι ήδη έχετε ξεκινήσει κάποια πιλωτικά προγράμματα. Ποια είναι η ανάλυση σας όμως για την κατάσταση της νέων και κοινής χρήσης. Υπήρχε πολιτική βούληση, τι θα συμβαίνει και ποιο ρόλο θα παίξει η δική σας υπηρεσία. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ορατότητα της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος σε αυτό το κεφάλαιο και τι μέσα θα χρησιμοποιήσετε από τη δική σας μεριά. Τέλος, για το θέμα των μη επανδρομένων οχημάτων. Να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο κ. Πάσκου. Θα διεξάγεται έρευνα για αυτά τα οχήματα και η έρευνα αυτή θα χρησιμοποιηθεί από το Horizon 2020, 2020 αν όχι από πού θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Λέζινγκ. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αρνού και όπως είπε και η κυρία Κρόνμπερ που μίλησε πριν από μένα θα με ενδιαφέρε να ακούσω μερικά παραπάνω πράγματα για την έρευνα που θα γίνει για τα μη επαδρομένα εναέρια οχήματα. Στις 19 Νοεμβρίου πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις ε, σχετικά. Εγώ ρωτώ τώρα, θα πρόκειται για μη επανδρομένα, μη εξοπλισμένα εναέρια οχήματα Αποκλείονται δηλαδή τα οχήματα που θα έχουν όπλα. Θα... Ε, επίσης, το αχρήματα για την έρευνα αυτή από πού θα προέλθουν από το δικό σας προϋπολογισμό της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ή από κάποιον άλλο προπολογισμό και ποια συγκεκριμένη τίτλο αυτού του άλλου προπολογισμού. Και άλλη μια ε, ερώτηση έχω για την έρευνα για αυτά τα ε, όπλα αν θέλετε ή τα ε, εργαλεία διτής χρήσης. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι να γίνουν αρκετά πράγματα για αυτά τα, τα αντικείμενα τα εργαλεία διτής χρήσης και εδώ πρέπει να γίνει μια κάποια έρευνα φαντάζομαι. Ε, ε, υπάρχει κάτι το πιο συγκεκριμένο και από πού θα προέλθουν τα χρήματα από τον ορίζοντα 2020 ή α, μήπως αυτό προσκρούει σε αυτό που λέγεται ότι θα, ε, η Ευρώπη δεν θα πρέπει να ασχολείται με οπλικά συστήματα κτλ. κτλ. Είναι αυτά τα 50 δις που αναφέρατε για τον προϋπολογισμό σας. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμετς. Σας ευχαριστούμε κύριε Αρνού που έρχεστε εδώ για άλλη μια φορά. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη είχαν και έχουν ένα καταπληκτικό κίνητρο αυτή τη στιγμή, ένα φοβερό ερέθισμα για να ασχοληθούν περισσότερο με το pooling and sharing, την συνένωση και κοινή χρήση και να καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν κοινού πόρους για κοινού στόχους. Λοιπόν, η κρίση είναι αυτό το φοβερό κίνητρο αυτή τη στιγμή, η οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση είναι ο παράγοντας αυτός ο οποίος ασκεί μια τεράστια πίεση και που ουσιαστικά υποκινεί τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συνένωση δυνάμεων. Ποια είναι η δική σας τώρα όμως η άποψη. Εγώ δεν βλέπω στην πράξη να έχει γίνει κάτι τέτοιο, να έχει λειτουργήσει το κίνητρο αυτό. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι λαμβάνονται αποφάσεις λανθασμένες, οι οποίες ουσιαστικά αντιτίθενται στην ε, προσπάθεια αυτή συνένωσης ε, δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, στη δική μου τη χώρα, είχαμε μία μονάδα παραγωγή ένα ναυπηγείο, το οποίο κατασκεύαζε σκάφη πλοία για, τη δική μας, την, για το δικό μας το πολεμικό ναυτικό, το πλοία τα οποία προφανώς χρειαζόμαστε εμείς για να προστατεύσουμε τη χώρα. Και βλέπουμε ότι αν τελικά δεν κατασκευαστούν αυτά στην Πορτογαλία θα πρέπει να τα αγοράσουμε από κάποια άλλη χώρα με όλες τις επιπλοκές που αυτό συνεπάγεται και με φαινόμενα διαφθοράς που πάρα πολλές φορές έχουμε σε τέτοιες αγορές. Η κυβέρνησή μας λοιπόν τι έκανε, κατέστρεψε, διέλυσε την αυπηγή αυτά και δεν έδωσε απολύτως καμία δικαιολόγηση γι' αυτό και αντιτάχθηκε βασικά και στην ίδια την γνώμη του πολεμικού ναυτικού και γενικότερα του στρατού. Ουσιαστικά τι βλέπουμε να γίνεται, ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο μας λέγατε εσείς ή που θα έπρεπε να κάνουμε. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μια ευρωπαϊκή τεχνολογική αμυντική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να εκμεταλλευόμαστε τι δυνατότητε που έχουμε και να συνεργαζόταν για παράδειγμα την ναυπηγείο τη Πορτογαλία με άλλα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, βλέπουμε να γίνεται το αντίθετο. Βασίζουμε λοιπόν στο παράδειγμα αυτό για να σα πω ότι χάσαμε μία πολύ σημαντική ευκαιρία. Θέλω επίση να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι εδώ στι Βρυξέλλες κάναμε τη δουλειά που θα έπρεπε να είχαμε κάνει αν έχουμε ανταποκριθεί στην αποστολή μας όσον αφορά τη διάρθρωση των διαφόρων υπηρεσίων, όχι μόνο στα πλαίσια του δικού σας του οργανισμού, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου υπάρχουν πολλές διευθύνσεις, οι οποίες ευθύνονται για τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμή μέχρι στιγμής και που δεν μας αφήνουν τελικά να φτάσουμε τους στόχους που έχετε θέσει τώρα όσον αφορά τα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βανόρντεν, εγώ δεν είμαι κατά της ανάπτυξης αυτών των αεροσκαφών και δεν είμαι κατά αυτής της τεχνολογίας. Θα ήταν πολύ σημαντικό όμω για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αλλά και για κάποια κοινοτικά προγράμματα όπως τον ορίζοντα 2020 να καταφέρουμε εκ των προτέρων να καθορίσουμε ποια θα είναι η χρήση των πορισμάτων αν θέλετε της έρευνάς μας εν προκειμένου των αεροσκαφών αυτών έτσι ώστε τα νέα τεχνολογικά αυτά μέσα να μην αντιταχθούν στο διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι ε, και ο δικός σας οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, θα πρέπει να επενθυμίσει την βασική αυτή ανησυχία στα κράτη-μέλη. Τέλος, αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα να συντοποιήσουν τα κράτη-μέλη το ότι ε, πρέπει να υποστηρίξουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα και να εκμεταλλευτούν τι νέε ευκαιρίε που απορρέουν από αυτόν. Τι κάνει όμω ο δικό σα οργανισμό γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε στελέχη βάθμα από διάφορες χώρες καταρτισμένα που να προέρχονται για παράδειγμα από το Υπουργείο Άμυνα ή από την αμυντική βιομηχανία και να συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι το μόνο τέτοιο άτομο από την Πορτογαλία έφυγε, αποχώρησε από, αυτό τον, από τον οργανισμό σας, τον απέλησαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό να διασφαλίσετε την διασύνδεση αυτή ανάμεσα στον οργανισμό σας και τα διάφορα κράτη-μέλη. Να μπορούν δηλαδή να αποτελούν τα σημεία επαφής, του συνομιλητές αν θέλετε, ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχουμε έναν τέτοιον εθνικό οργανισμό, αρμόδιο για, την, για τους αμυντικούς εξοπλισμούς, ο οποίος θα μπορούσε να αποφεληθεί βέβαια αν υπήρχε ένας Πορτογάλος στο δικό σου οργανισμό που ήταν σε θέση να ενημερώνει τον δικό μας τον οργανισμό. Η κυρία Παναγιώτοβα έχει το λόγο, σύντομα παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομη, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αρνού, ποια είναι η προσωπική σας άποψη όσον αφορά την ιδέα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού εξαμήνου άμυνας για να καταφέρουμε να εξορθολογήσουμε τους εθνικούς αμυντικούς προπολογισμούς. Θα αποτελέσει αυτό προστιθέμενη αξία για το δικό σας τον οργανισμό. Θα δώσει μια νέα ευκαιρία στο δικό σας τον οργανισμό όπως ακριβώς δίνει νέες ευκαιρίες πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αρνού, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ορισμένες δεν είναι εύκολες. Πρώτα πρώτα λοιπόν για την ερώτηση του Προέδρου για τον προπολογισμό του οργανισμού μας. Ε, είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Έχουμε ένα σωρό ναι, καθήκοντα και νέες εντολές που μας ανατίθενται και υπάρχει και συγχρόμη μείωση του προπολογισμού μας. Ε, Απ' την άλλη μεριά τα νίκια δεν πέφτουν, τα πάγια έξοδα δεν πέφτουν και πραγματικά έχουμε μειωμένο προϋπολογισμό με αύξηση των καθηκόντων μας. Γιατί διότι ο προπολογισμό περνάει με ομοφωνία. Δεν υπάρχει ομοφωνία για να δοθούν παραπάνω χρήματα. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε ορισμένες ε, δραστηριότητες να τις αναβάλουμε για το μέλλον. Τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, το ΣΕΖΑΡ παραδείγματος χάρη που είναι ad hoc δραστηριότητες τα αναβάλουμε ή τα αντιμετωπίζουμε με μικρό αριθμό ατόμων. Προσπαθούμε να δούμε βεβαίως τα αμυντικά προ, προ, από αμυντική άποψη τα θέματα ε, που εντάσσονται στο ΣΕΖΑΡ και να τα αντιμετωπίσουμε. Τέλος πάντων δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλα αντίστοιχα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είσαστε στο Μόναχο, οι περισσότεροι από εσά αν υπάρχουν καινούργιε ιδέες, καινοτόμες ιδέες για τον προπολογισμό του οργανισμού ε, είναι ευπρόσδεκτες. Τώρα τα πράγματα είναι όπως είναι, βρέχει πρόθεσμα, δεν πρόκειται να αλλάξει κατάσταση. Ε, μακροπρόθεσμα μπορεί, αλλά η επιλογή ορισμένων ad hoc δράσεων ε, μου φαίνεται καλή ιδέα. Τι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα βέβαια και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε εμά δουλεύουν παραπάνω ε, αλλά τουλάχιστον δουλεύουν. Ελπίζω πάντως ε, πέρα από αυτές τις ε, δράσεις ad hoc να μπορέσουμε να βρούμε και άλλα μέσα για να μπορέσει να επιζήσει ο οργανισμός μας. Τώρα για τις συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες. Ναι, έχουμε επαφές με τις τρίτες χώρες που αναφέρατε, τις ε, ανατολικής εταιρικής ε, έτσι κι αλλιώς με την Νορβηγία, την Ελβετία και τη Σερβία πρόσφατα είχαμε διοικητικές ε, επαφές. Αλλά ε, η Γεωργία μας επισκέφθηκε σε υψηλό επίπεδο, η Ουκρανία ήρθε σε επαφή μαζί μας και η Ρωσία και όλο και περισσότερο έρχονται τρίτες χώρες και, και δηλώνουν το ενδιαφέρον τους. Ε, η Ιαπωνία και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα η Γεωργία και η Ουκρανία έχουν ήδη πάρει κάποιες ε, κάποια σχέδια ε, προγραμμάτων και είναι δικό τους θέμα αν θα υπογράψουν ή όχι. Τώρα για αυτό που είπε ο κύριος Πασκού δεν ξέρω τι θα γίνει στο Συμβούλιο της, του οργανισμού μας, κατά πόσον θα έρθουν οι Υπουργοί Εκοφήν στο Συμβούλιο μας. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα χρειάζεται να κάνουμε μια συζήτηση ε, που στην οποία να εμπλακούν και Υπουργοί Οικονομικών. Δεν γίνεται να ανταποκριθούμε στις αρμοδιότητες που μας ανατέθηκαν, τις εντολές που μας δόθηκαν με τον προπολογισμό που έχουμε. Ελπίζουμε, ε, μάλλον οι Υπουργοί Εκοφήν έτσι κι αλλιώς έχουν εντολές από τους αρχηγούς και ε, κρατών και κυβερνήσεων ε, αντίστοιχες με αυτές που παίρνουμε κι εμείς. Όταν αυτά που λένε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν αφορούν τον καθένα χωριστά, αφορούν όλους μας μαζί. Όταν μας αναθέτουν λοιπόν κάποιες εντολές ως οργανισμό άμυνας θα πρέπει και ο, τα αντίστοιχα Υπουργεία Οικονομικών να κάνουν ε, και, αυτό, αυτό, και αυτά αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έγινε η μεγάλη στροφή 180 μοιρών που ρωτήσατε τι να πω, εγώ δεν είμαι ε, ειδική στην οδήγηση σε διάφορες χώρες αλλά όταν ανεβαίνει κανείς μια ανηφόρα ε, βάζει μεγάλη επιτάχυνση στην αρχή νομίζω ότι αυτή η επιτάχυνση δόθηκε αυτή τη στιγμή και η μηχανή άρχισε να προχωρεί Τώρα, για τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα, θα τα χρησιμοποιήσουμε για τη στρατηγική μας για την προστασία των θαλασσών, ασφάλεια των θαλασσών. Η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, παρατη, θα χρησιμοποιηθούν drones ως παρατηρητήρια για τις θάλασσες και αυτό θα συζητηθεί. Τώρα, για το θέμα της συνένωσης και κοινή χρήση, το pooling and sharing που η κυρία Κρόνενμπερκ, προτείναμε ένα ε, κώδικα δεοντολογίας που υπέ, για το θέμα αυτό που... Ε, έγινε δεκτός από τους υπουργού Άμυνας των ε, κρατών μελών και τώρα πρέπει να δούμε να κάνουμε την αξιολόγησή μας. Μετά από ένα χρόνο που θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση δεν ξέρω αν θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι θα δούμε τι έχει γίνει και πού μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Τι να ε, θα δούμε ξανά το πλαίσιο πολιτικής, τα κίνητρα κτλ. Για να ξεπεράσουμε το 14, γιατί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καταλάβαμε ότι πρέπει να πάμε πέρα από τον κώδικα αυτό ε, δεοντολογίας και η ιστορία αυτή της αξιολόγησης είναι πραγματικά ε, πρόκληση την οποία όμως θα αντιμετωπίσουμε. Τώρα όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα, την ορατότητά μας, την παρουσία μας, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Με τα χρήματα που είχαμε στη διάθεσή μας αναλάβαμε δράσεις επικοινωνίας ε, και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήρθαμε σε επαφή με τον πρόεδρο, με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης κλπ για να φτιάξουμε ένα κοινό ανακοινοθέν και δώσαμε και υλικό για αυτό το ανακοινοθέν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε να πάμε παραπέρα. Αν πάω εγώ σε μία συνέντευξη τύπου ως εκπρόσωπος του οργανισμού άμυνας ε, εντάξει, καλό είναι αυτό, ήδη είναι καλό και θα πιστεί όποιος πιστεί. Τώρα άμα όμως έρθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έρθει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έρθουν τα κράτη-μέλη και πούν κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά, αυτό βεβαίως έχει μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο, είναι κοινωνιακά πιο καλό και πιο μεγάλο. περιμένουμε ότι τώρα η αιρετή πολιτική, οι κυβερνήσει των κρατών μελών είναι αυτοί που πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία μας αν θέλετε και την ορατότητά μας. Τώρα για την έρευνα και τα drones. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά σκέλη έρευνας. Εμείς επικεντρωνόμαστε πρώτα-πρώτα σε εκείνα τα θέματα που έχουν διπλή χρήση. Έτσι, ε, για ε, εργαλεία αν θέλετε τα οποία μπορούν να μπουν και στον κανονικό εναέριο χώρο ως τον ειδικό εναέριο χώρο που είναι περιορισμένος για στρατιωτικά ε, οχήματα. Λοιπόν, ε, και γι' αυτό αναφέρθηκα άλλωστε και στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό πριν και στο Σεζάρ και είπαμε ότι επιλέξαμε ορισμένα πράγματα εκεί. Τα κράτη-μέλη ήδη έχουν δεσμεύσει 50 εκατομμύρια για τον για το θέμα αυτό από τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης για τα, εργαλεία, αν θέλετε, τα μέσα διητής χρήσης, στρατιωτικής και μη στρατιωτικής. Για τις ε, στρατιωτικές δυνατότητες τώρα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, μίλησαν για επιτήρηση και εποπτεία. Ε, όπως είπε και ο τέραρχος Ρουσιέ δεν πρόκειται να αναλάβει στρατιωτικός το ο, πιλότος το πιλοτάρισμα του ο, πιλότος μαχητικού την, το πιλοτάρισμα του drone ε, εκεί θα πρέπει να προσέξουμε βέβαια όπως ξέρετε εδώ πρόκειται σε τελευταία ανάλυση για αποφάσεις των κρατών μελών που μέσα στα πλαίσια των εσωτερικών τους δομών θα πρέπει να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Νομίζω ότι υπήρξε μια παρεξήγηση κάποια στιγμή. Δεν θα δημιουργηθεί δύναμη ευρωπαϊκή ε, δύναμη drones. Ε, ε, ε, για τη νέα γενιά drones για παρατήρηση βεβαίως θα γίνει δουλειά διότι εκεί μιλάμε για διπλή χρήση όπως σας είπαμε πολιτική και στρατηγική τη στρατιωτική. Εκεί βέβαια θα, η χρηματοδότηση εν μέρη θα προέρθει από τον ορίζοντα 2020, όχι όμως αποκλειστικά. Η κυρία Κόμες αναφέρθηκε στην κρίση που βιώνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Όντως είναι λίγο αμφιλεγόμενος ο ρόλος της κρίσης. Ε, ξεκίνησε η κρίση ορισμένα πράγματα δεν υπάρχει ε, βέβαια εναλλακτική λύση η μόνη εναλλακτική θα ήταν να καθίσουμε σταυρωμένα χέρια και να σκοτώσουμε τη βιομηχανία μας τελικά τη στρατιωτική μας βιομηχανία ε, και ε, δεν θα υπάρχει και δρόμος επιστροφής αν κάνουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αλλά γιατί εμείς επιμένουμε τόσο πολύ στα προγράμματα, χρειαζόμαστε προγράμματα ούτω ώστε η βιομηχανία όπλων μας, η βιομηχανία μας να έχει συγκεκριμένες διορίες, προθεσμίες και να ξέρει πολύ συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνει διαφορετικά δεν μπορεί να δικαιολογήσει και τις επενδύσεις της η βιομηχανία των κρατών μελών. Τώρα αναφερθήκατε και κάτι τι άλλο δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τα ναυπηγεία τα πορτογαλικά όπως ξέρετε κανείς και από εκεί και πέρα για την συμμετοχή της Πορτογαλίας στο, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας κανείς δεν απολύθηκε ε. Α, αλλά άμα λήξει το συμβόλαιο του πάβει να είναι υπάλληλο του οργανισμού και, αλλά μπορεί να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα για άλλη θέση. Τώρα, ε, επίσης, ε, ε, έχουμε 120 θέσεις μόνο ε, και προσπαθούμε να επιλέξουμε τους καλύτερους για, το, για αυτές τις 120 θέσεις με ειδικέ γνώσεις για ε, ε, να ανταποκριθούμε στις εντολές που μας δόθηκαν. Ε άνθρωποι αυτοί είναι στην υπηρεσία των κρατών μελών δεν εκπροσωπούν όμως και δεν συμφωνώ με την ορολογία αυτή ότι εκπροσωπούν και είναι αντιπρόσωποι κάποιου κράτους μέλους Επουδενή ε, δεν λόγο τώρα για το ευρωπαϊκό εξάμεινο η κάθε Άνστον στο πρόγραμμα της ε, είπε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο θα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σίγουρα δεν μπορεί να είναι ε, το ακριβές αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού αντίγραφο του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε κάτι ε, αντίστοιχο και μέσα στο θεσμικό να δούμε το θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών, το ρόλο των κοινοβουλίων για θέματα άμυνας και μετά να βρούμε μια κάποια ισορροπία για να κάνουμε κάτι το οποίο θα ήταν στη τελευταία ανάλυση στον τομέα της άμυνας κάτι συμπληρωματικό προς το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ πυκνή, πυκνές οι απαντήσεις σας, πολύ ακριβείς όπως κάθε φορά. Δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να τα ξαναπούμε πριν να ξεκινήσει η επόμενη θητεία. Το ίδιο με τον κύριο Ρουζιέ. Ευχαριστούμε πολύ και για την υποδοχή που μας επιφυλάξατε στην ίδια την υπηρεσία είναι σημαντική, σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ορατότητα της. Γι' αυτό το λόγο πήγαμε εκεί με κάποιους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή. Ήταν πολύ χρήσιμη η επίσκεψή μας. Συνάδελφοι μου εξέφρασαν τόσο την ικανοποίησή τους όσο και το γεγονός ότι δεν ήξεραν τι ακριβώς κάνει η υπηρεσία σας νωρίτερα ιδιαίτερα για παράδειγμα για τον ενιαίο ουρανό. Το έργο σας είναι εξαιρετικά χρήσιμο και είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τους ε, ευρωβουλευτές όσο και τους ε, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η συνάλφοι στην επόμενη θητεία αλλά και η συνάλφοι στα Εθνικά Κοινοβούλια ελπίζω ότι θα σας ξαναεπισκεφτούν. Και θα συναντήσουν τους ανθρώπους που θα είναι υπεύθυνοι ιδιαίτερως για την ε, ε, προώθηση των θεμάτων τα οποία σας ανέθεσε το Συμβούλιο Κορυφής. Για τα διάφορα άλλα τα οποία <laughs> είπατε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ε, θα δούμε στα ενδιάμεσα στάδια πώς πηγαίνει η δουλειά. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και να συνδιαλεγόμαστε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια περί του ρόλου του Κοινοβουλίου και της δικής μας Επιτροπής σε ό,τι αφορά το πώς επηρεάσαμε κατά κάποιο τρόπο τις εργασίες του Συμβουλίου. Η ανταλλαγή πληροφοριών για τα πολύ τεχνικά θέματα της υπηρεσία σας είναι πολύ σημαντική. Η πολιτικοποίηση με την καλή έννοια του όρου των τεχνικών ζητημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς ως Ευρωβουλή ε, συνδέουμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες και την κοινή γνώμη. Λοιπόν, θέματα τα οποία είναι πολύ τεχνικά και συγκεκριμένα, ίσως είναι χρήσιμο να τα βλέπουμε εμείς από πολιτικής και στρατηγικής πλευράς μέσω των συζητήσεων που γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Γιατί σας περιμένει πολλή δουλειά τον επόμενο 1,5 χρόνο. Ε, ε, διακοπή για ένα λεπτό για να χαιρετήσουμε την κυρία Αρνού και ξεκινάμε την κοινή συνεδρία, α το πούμε έτσι, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ΣΕΝΤΕ. Euh, chers collègues, mesdames, messieurs. <laughs> nous avons minutes devant nous. Ωραία. Κυρίε και κύριοι, έχουμε 20 ακόμα λεπτά στη διάθεσή μα. Θα είμαστε γρήγοροι. Πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤΣΕΝΤΕ για να κάνουμε τη συζήτηση που δεν κάναμε στην ΑΦΕΤ για το θέμα της έκθεσης για την συνολική προσέγγιση. Έχουμε εδώ τον κύριο Πάσκου, αντιπρόεδρο της ΑΦΕΤ, στον οποίο δίνω το λόγο. Ας συνεχίσουμε να αυτοσχεδιάζουμε. Είναι η δεύτερη εξέταση της ολιστικής προσέγγισης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, ε, των επιπτώσεών της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο προσχέδιο το είχατε πάρει, το είδατε, υποβάλατε 76 τροπολογίε Στην περασμένη εβδομάδα στο Τρασβούρο είναι μια συνάντηση με του πιο ηγητέ, ορισμένοι εξ αυτών είναι παρόντε. Οπότε νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα σα δώσω το λόγο για να μα παρουσιάσετε την έκθεσή σα. Θα είμαι συντομότατο, λέει ο κ. Να ευχαριστήσω καταρχήν του και που εμπλούτησαν την έκθεσή μου, υπέβαλαν τροπολογίες και όχι μόνο αυτή βέβαια, χωρίς να την υπερφορτώσουν. Το θέμα είναι πολύ πλατή, έχουμε, μιλάμε για την ολιστική προσέγγιση, διατρέχαμε τον κίνδυνο ε, να διασπαστούμε ε, σε ό,τι αφορά το, τα μηνύματά μας. Το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι η ανάγκη συντονισμού. Η ολιστική προσέγγιση είναι ε, προφανώς ε, εύλογη φιλοδοξία και αξιέπαινη ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αμφισβητούμε που είναι ότι θα πρέπει να είναι στόχος μας. Από την άλλη μεριά η έκθεση ε, εντοπίζει ένα αριθμό όχι δυσλειτουργιών αλλά τουλάχιστον αδυναμιών ή περιορισμών της ολιστικής προσέγγισης έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Ε, έχουμε ακούσει πολλά λόγια, πολύ ρητορική αλλά η ολιστική προσέγγιση απαιτεί στην πραγματικότητα εξαιρετικό συντονισμό ανάμεσα στα μέσα που διαθέτει η Κομισιόν, την Επιτροπή Εξωτερική Δράση, ορισμένε φορέ τα κράτη-μέλη, ορισμένε φορέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο συντονισμό αυτό θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα, εκ των προτέρων και αυτή τη στιγμή χωλαίνει. Και αν πάμε ακόμα πιο μακριά στη σκέψη μας, η ολιστική προσέγγιση πολύ συχνά επενείται από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των υστέρων. πολλές φορές η, ε, η ε, μας λέει για παράδειγμα ε, θέσαμε σε εφαρμογή την ολιστική προσέγγιση στο κέρας Αφρικής αλλά αυτό εκ των υστέρων μας το λένε δεν υπήρχε μια εκ των προτέρων στρατηγική συντονισμού γι' αυτό το λόγο ασφαλώς χρειάζεται η ανάπτυξη του συντονισμού μεταξύ όλων των μέσων που μπορούν να κινητοποιηθούν αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διαθέτουμε και ε, στρατηγικές εκ των προτέρων, στρατηγικές, ε, περιφερειακές στρατηγικές. Όπως για παράδειγμα για το Σάχελ. Ε, ε, μια στρατηγική για τις θάλασσες, για τη θαλάσσια ασφάλεια κλπ. Αυτά θίγω στην έκθεσή μου. Και πάλι δεν έχουμε σημαντικές ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ομάδες Επιμένουμε σε ό,τι αφορά την ε, ανθρωπιστική πολιτική και την αναπτυξιακή πολιτική, πολύ σημαντικά κομμάτια της ολικής προσέγγισης. Το ευαίσθητο σημείο βέβαια μπορεί να είναι το διαφορετικό πολιτικό στάτους των ιδιαίτερα των ανθρωπιστικών εργαλείων που διαθέτουμε αφενός και των εργα... στρατιωτικών εργαλείων από την άλλη μεριά. Τα ανθρωπιστικά εργαλεία, τα ανθρωπιστικά μέσα που διαθέτουμε, ιδιαίτερος η ΕΚΟ, ε, ε, ε, είναι ε, επιθυμούν διακαώς να διατηρήσουν την αυτονομία τους. Ε, αυτή η αυτονομία τους εξασφαλίζει την ουδετερότητά τους ε, και την πρόσβαση παντού εκεί όπου δρούν. Παρόλα αυτά, όλη αυτή η δράση ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτείται από, τα όργανα της Ευρωπαϊκής, από τον προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολιτικά όργανα. Οπότε, ναι, σεβασμό στην ανεξαρτησία, την καθολικότητα της ανθρωπιστικής δράσης, την ουδετερότητα, αλλά χρειάζεται συντονισμός. Συντονισμός εκ των προτέρων ε, και με, με αυτό το συντονισμό μειώνουμε τον κίνδυνο χασμοδιών ε, ή αδυναμιών τη στιγμή που θα ε, δράσουμε. Ο συντονισμός βέβαια θα πρέπει να γίνεται και επί τόπου και στο θέατρο των επιχείρησεών μας, εκεί θα πρέπει να συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε, δηλαδή θα περιοριστούμε μόνο στον εκ των προτέρων συντονισμό. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της έκθεσης. Ευχαριστώ και πάλι τους ε, συναδέλφους που υπέβαλαν αυτές οι 78 τροπολογίες. Έχουμε 8 συμφωνίες ε, ε, σε συμβαστικές προτάσεις, αυτό είναι την εβδομάδα. Υπέβαλα άλλη μία πρόταση συμβασμού σε σχέση με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών που ήταν αρκετά μακροσκελής, ε, πιο μακροσκελής και από την ίδια, από την ίδια έκθεση. Οπότε υποβάλλω, υπέβαλα μια συμβαστική τροπολογία που περιλαμβάνει βασικά ε, τις βασικούς άξονες της γνωμοδότησης Επιτροπής Γυναικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όντω δεν μπορούμε να μιλάμε για ολιστική προσέγγιση χωρίς να υπάρχει μία εκ των προτέρων στρατηγική θα ξέρετε ότι το να συγκεντρώνουμε απλώς τα διάφορα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση δεν αρκεί για να έχουμε πραγματικά ολιστική προσέγγιση. Μαρία Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρετε ότι ε, ζούμε σε ένα κόσμο όπου τα σύνορα είναι λίγο πιο, όλο και περισσότερο πιο ασαφή ανάμεσα σε αυτό που αποτελεί εσωτερικό και εξωτερικό τελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται συνεκτικότητα όχι μόνο θεσμική αλλά και πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι ο κατακαιρματισμός της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά αποτελεί πολύ μεγάλη αδυναμία για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θέλει να γίνει παράγοντας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση, η οποία να περιλαμβάνει όμως και μια κάποια συνεκτικότητα, μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική που ακολουθούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την πολιτική που ακολουθούν μονομένα τα κράτη-μέλη για πολλούς τομείς εσωτερικά και εξωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά την πολιτική απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει να μας απασχολούν μόνο οι εξωτερικές σχέσεις γενικά και αόριστα, αλλά και οι σχέσεις που έχουμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη, οπουδήποτε ουσιαστικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τοποθετηθούμε πολιτικά. Η έκθεση λοιπόν αυτή νομίζω ότι θα πρέπει να διευρυνθεί περισσότερο και να γίνει πιο συγκεκριμένη σε κάποια σημεία. Ξέρω το εγχείρημα είναι δύσκολο γιατί το ίδιο το θέμα είναι πολύ φιλόδοξο. Οι σοσιαλιστές υπέβαλαν λοιπόν πολλές τροπολογίες για να βελτιώσουν και να καταστήσουν πιο συγκεκριμένη την τόσο ευρία και γενική αυτή έκθεση. Νομίζουμε πάντως ότι με τις τροπολογίες αυτές που έχουν κατατεθεί εν μη τι άλλο διευκρινίζονται δύο πράγματα. Ποια είναι καταρχάς η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε, λέμε στις τροπολογίες μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσει κάποιες αρμοδιότητες που έχει στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής, όπως έγινε για παράδειγμα τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις αρμοδιότητες που έχουμε στην εξωτερική πολιτική και αυτές οι αρμοδιότητες να συντονίζονται με αρμοδιότητες που έχουμε σε άλλες πολιτικές, όπως για παράδειγμα στην ενεργειακή πολιτική. Ξέρετε ότι ε, το πολύ ψηλό κόστος της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυναμώνει τελικά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και για ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Αποδυναμώνει τη σχέση μας με τους άλλους εταίρους. Νομίζω λοιπόν ότι το μήνυμα αυτό θα πρέπει να φτάσει στην ε, αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον εισηγητή, τον κύριο Ντανζό. Έχουμε προτιμάσει εμείς τον κατάλογο ψηφοφοριών και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή για την επικοδομητική συνεργασία που είχε με τους κοιόδη εισηγητές. Ευχαριστούμε κυρία Λέζιν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα φαντάζεστε βέβαια ότι η πολιτική μου ομάδα έχει σοβαρές ε, διαφωνίες όσον αφορά ε, τη βασική φιλοσοφία θα υποβάλω μια έκθεση μειοψηφίας το λέω ήδη από τώρα και θα το εξηγήσω λοιπόν πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω για τα πολύ ξεκάθαρα πράγματα που είπε ε, που λέει εδώ ο εισηγητής η σαφήνεια που επιδεικνύει για, τη, για την ε, ε, για έναν <laughs> κόσμο που μεταλλάσσεται ε, και πώς αλλάζουν τα πράγματα και τα λοιπά. Ωραία, μέχρι εκεί είναι σαφές. Αλλά εγώ θα το έκανα ακόμη πιο σαφές μιλώντας για αλλαγή γεωστρατηγικών ισορροπιών ε, και αυτό δεν αναφέρεται ιδιαίτερα στην έκθεση. Σε κάποιο άλλο σημείο τι σημαίνει ακριβώς ε, πολυ, θέματα εσωτερικής πολιτικής που επηρεάζουν όμως την εξωτερική πολιτική. Τι θα πει αυτό. Αυτό με ανησυχεί σφόδρα είναι προφανές ότι ότι για τα θέματα ε, της χρηματοδότησης και για χρησιμοποίηση ας πούμε απόρων τύπου ε, Αφρικής για στρατιωτικούς σκοπούς αυτό για την ε, ειρήνη στην Αφρική που υπάρχουν κάποια κονδύλια να τα βάζουμε εδώ για στρατιωτικούς σκοπούς ε, αυτά μας βρίσκουν αντίθετους και όσον αφορά και για τη διτή σχέση στρατιωτικού και μη στρατιωτικού ε, για τους φορείς αυτούς διτής ε, προσέγγισης στρατιωτικής και μη στρατιωτικής αυτό εδώ υπάρχει μια σύγχυση κύριε Ντόνζο και θα θέλαμε να το τονίσουμε επίσης σε κάποιο σημείο περιγράφεται την αναγκαιότητα για την ουδετερότητα κάποιων πολιτικών δράσεων και από την άλλη μεριά μιλάτε για την ε, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων όπου ουσιαστικά επιβάλλει κάποιους πολιτικούς κανόνες. Λοιπόν τι γίνεται, ουδετερότητα ή όχι. Ε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια κάποια σύγχυση. Επίσης αναφέρεται συνεχώς η ταχύτητα ή βιασύνη και αυτά πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα και βιαστικά για να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Συγγνώμη, τα κράτη-μέλη μπορεί να έχουν ορισμένα προγράμματα τα οποία οποία ε, είναι και στρατιωτικά και μη στρατιωγή. Στρατιωτικά μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να παρθούν αποφάσεις. Έχω την εντύπωση ότι αυτά που λέτε εδώ ουσιαστικά ε, θέτουν σοβαρά ερωτήματα για τις δημοκρατίες μας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε την κυρία Μινής ε, για την εργασία που έκανε. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε, όπως το είπατε και εσείς, πολύ επικοδομητικά για ένα πολύ ευρύ θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προφανώς θέλουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ στόχος τελικά είναι να εμπλουτιστεί η έκθεση αυτή, η οποία προσπαθεί ουσιαστικά να υιοθετήσει κάποιες βασικές κατευθύνσεις. Να εμπλουτίσουμε χωρίς να υπερφορτώσουμε την έκθεση αυτή. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε όλοι και αυτό κάνετε και εσείς με τις τροπολογίες σας για κάποιες ενδεχομένως να υποδείξω αρνητική ψηφοφορία γιατί υπερβαίνουν ένα κάποιο βαθμό λεπτομέρειας. Επί της αρχής και επί της ουσίας δεν αντιτίθεμαι σε αυτές τις τροπολογίες αλλά νομίζω ότι εμπεριέχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και μπούμε σε τόσες πολλές λεπτομέρειες για επιμέρους σημεία, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό για όλα τα υπόλοιπα και τότε κινδυνεύει να μην είναι πολύ καλή έκθεση. Κύριε Λέζινγκ, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Αναφέρεστε σε κάποια ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν από την αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας, κυρίως για την διάρθρωση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας. Εμείς στην έκθεση αυτή εγώ μάλλον στην έκθεση αυτή, θέλησα να καταγράψω τι έχει συμβεί από την συνθήκη της Λισαβόνας και μετά και από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή πολιτική εξωτερική πιο ισχυρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς όμως να θέσουμε ένα αμφιβόλο τις αρχές οι οποίες διέπουν όλες τις ανθρωπιστικές αποστολές που διέπουν βασικά τη δράση οποιασδήποτε μη κυβερνητικής ή κυβερνητικής οργάνωσης. Ουσιαστικά θέλουμε να ακολουθούμε πάντα την αρχή της ουδετερότητας. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, εντάσεις αλλά δεν νομίζω ότι είναι αντιφατικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή για κάποιες εμπόλεμες ζώνες και παράλληλα να έχει κάποια μέσα που θα επιτρέπουν στην Ένωση να βοηθήσει όλους τους κατοίκους των περιοχών αυτών ανεξάρτητα με την πολιτική θέση που έχει ε, εγκρίνει. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να τηρήσουμε αυτή την διαχωριστική γραμμή, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τώρα, αναφερθήκατε σε κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει ανέκαθεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις διάφορες κρίσεις. Στις ε, συζητήσεις που μόλις τώρα κάναμε με τον κύριο Ντερουζιέ και με την ε, κυρία Αναγκόμες μάλλον πήρε το λόγο και είπε ότι ε, πολύ συχνά οι ίδιοι στρατιωτικοί δεν μπορούν να αποφανθούν για την αποστολή στην Λιβύη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μη στρατιωτική. Αυτό προφανώς επηρεάζει την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία, αλλά ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σαφής οριοθέτηση αρμοδιοτήτων. Οι πολιτικά ευθύνοντες δεν μπαίνουν στον τομέα το στρατιωτικό και οι στρατιωτικοί με τη σειρά τους δεν εμπλέκονται στα μη στρατιωτικά θέματα. Ξέρω ότι Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε την εξή κατάσταση. Πολλέ φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διαχείριση κάποιων κρίσεων φτάνει μετά τη μάχη όπως λέμε στα γαλλικά. Ουσιαστικά επεμβαίνει εκ των υστέρων πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα. Η κινητοποίηση λοιπόν των δυνατοτήτων της είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, πολλές φορές είναι πολύ πολύπλοκη υπόκειται πάρα πολύ συχνά στην καλή πολιτική βούληση των κρατών μελών, όπως για παράδειγμα είδαμε στην τελευταία αυτή αποστολή, όπου έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια ανθρωπιστική κρίση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Βλέπαμε εκ των προτέρων ότι ερχόντουσαν, υλοποιόντουσαν σιγά σιγά διάφορα καταστροφικά σενάρια, γίνανε συζητήσεις στα Ηνωμένα Έθνη, ο κύριος Ντερουζιέ μας το είπε ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Μάρτιο για να δούμε μια πραγματική ευρωπαϊκή δύναμη επιτόπου, ενώ για παράδειγμα οι Γάλλοι ανέλαβαν δράση ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου. Πάντως συμφωνώ μαζί σας σε ένα σημείο. Πολλές φορές ε, δεν προτρέχουμε ακριβώς, αλλά υπάρχει μια κάποια σύγχυση κατά την κινητοποίηση των διαφόρων δυνατοτήτων. Υπάρχουν ε, οι διάφορες γενικές διευθύνσεις, ΔΕΦΚΟ και άλλες ε, που ασχολούνται κυρίως με τα ανθρωπιστικά ζητήματα που θα κινητοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα, άλλες πάλι διευθύνσεις οι οποίες θα κινητοποιηθούν με μια κάποια καθυστέρηση και όντως δεν υπάρχει αυτός ο ευκταίος συντονισμός. Σαφώς λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα αυτό μέσω ενός πολύ πιο στενού και ισχυρού συντονισμού. Πάντως σε καμία περίπτωση εγώ δεν είπα και δεν λέω στην εκθεσή μου αυτή ότι υπάγεται ο ένας τομέας των άλλων. Ότι για παράδειγμα ο μη στρατοτικός τομέας πρέπει να υπαχθεί στο στρατοτικό ή το αντίστροφο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, ένας κίνδυνος στρατικοποίησης των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στρατό είναι ο στρατό, είναι εκεί πέρα που πρέπει να βρίσκεται. Απευθυνόμαστε σε αυτόν για να μα βοηθήσει όποτε το χρειαζόμαστε, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία στρατιωτικών και μη στρατιωτικών πτυχών και συνιστοσών σε διάφορε αποστολέ. Όπω είπε και η κυρία Μινής, στον παγκοσμιοποιημένο αυτό κόσμο τον οποίο, στον οποίο ζούμε, οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνουμε εμείς για την εσωτερική μας οργάνωση έχει επίπτωση στο μήνυμα το οποίο στέλνουμε, στέλνουμε εξωτερικά. Η διοργάνωση, για παράδειγμα, της εσωτερικής μας αγοράς προφανώς έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε την εμπορική μας πολιτική, η οποία αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εξωτερικής μας πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν είναι αρκετά ευρωπαϊκή ακόμα, δεν είναι αρκετά συλλογική. Βλέπουμε όμως ότι η παραμικρή απόφαση ή σχέδιο απόφασης που λαμβάνεται όσον αφορά την πολιτική ασύλου, όσον αφορά την πολιτική κυκλοφορία των πολιτών, ανθρώπων, μάλλον τρίτων χωρών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς επηρεάζει τις σχέσεις μας με τις χώρες της, ε, του Νότου τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα περισσότερα μεταναστευτικά ρεύματα. Προφανώς λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εσωτερική και την ε, εξωτερική πολιτική μας η οποία ακόμα προφανώς δεν είναι πλήρης. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι το ένα όμως επηρεάζει το άλλο. Αποφάσεις εσωτερικής πολιτικής επηρεάζουν για παράδειγμα τις σχέσεις που έχουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Υπάρχει λοιπόν μια αλληλοεξάρτηση ανάμεσα στις εσωτερικές και την εξωτερική μας πολιτική. Και έχετε προφανώς δίκιο ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο ακριβείς για τα σημεία αυτά στην έκθεση και όντως να ζητήσουμε να αποσαφινιστούν κάπως τα πράγματα. Δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνο για ποια αρμοδιότητα τελικά όταν μία απόφαση εσωτερική επηρεάζει τελικά την εξωτερική μας πολιτική ευθύνεται εν τέλει κάποιος επίτροπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτός είναι ο τελικός αρμόδιος, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Νομίζω το ερώτημα αυτό πρέπει όντως να το θέσουμε. Στο πεδίο εφαρμογή όμω και στο πλαίσιο τη επεξεργασία αυτή τη έκθεση ήταν πολύ δύσκολο να αποσαφηνίσουμε όλα αυτά τα σημεία. Εγώ θέλω να ακολουθήσουμε απλώ κάποιου γενικού προσανατολισμού και ας μην ξεχνάμε ότι η ιδιαιτερότητα του ζητήματος αυτού έγκυται στο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η περίφημη αυτή ολιστική προσέγγιση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Τα μέσα τα οποία σχολιάζουμε στην έκθεση αυτή βρίσκονται ακόμα υποκατασκευή, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης, που είναι μια υπηρεσία πολύ νέα. Πρέπει να ξέρετε ότι για μια πολιτική ασφάλειας και άμυνας, το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε δεκαετία ή μόνο πέντε χρόνια για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι χρονικά διαστήματα πάρα πολύ σύντομα. Ξέρετε ότι οι διπλωματικές υπηρεσίες στα κράτη μας έχουν ιστορία αιώνων. Αυτό λοιπόν ακριβώς προσπαθώ να κάνω στην έκθεση, να τονίσουμε όλα αυτά τα σημεία, τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσουμε απλώς κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. <laughs> Ε, ολοκληρώθηκε προφανώς η ε, συνεδρίαση της ΑΦΕΤ. Η ΣΕΝΤΕ θα ξανασυνεδριάσει εκτός μικροφώνου πρόεδρος.